Σας καλωσορίζω. Καλωσορίζω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτολή, Επιτροπή και θα δώσω τον λόγο στα δύο αυτά όργανα σε λίγο. Έχουμε την κοινή συζήτηση για τους μηχανισμούς ενίσχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης. Έχουμε μια δήλωση του Συμβούλιο διότι θα μας μιλήσει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της 7ης Μαΐου 2010. Θα έχουμε επίσης προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στη στρατηγική ΕΕ 2020 και τη διακυβέρνησή της και προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τη σημασία της στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ο πρώτος ομιλήτης εξ ονόματος του Συμβουλίου δίνω τον λόγο στον ε, κύριο Καριντά, υφυπουργό. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι διανύουμε μία περίοδο ε, εξαιρετικών και ε, οικονομικών αναταραχών. Πριν από λίγους μήνες ε, ξεκίνησε αυτή η κρίση και ε, μάλιστα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια περίπου όταν υπήρξε η κρίση των subprimes στις Ηνωμένε Πολιτείες. Άρα λοιπόν αυτή ε, η κρίση ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κρίση στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα και ε, γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι το οποίο επιδρά στην πραγματική οικονομία με τη μορφή μιας βαθιάς ύφεσης ύφεση λοιπόν ε, και όπου μειώθηκε η παραγωγικότητα και αυξήθηκε σημαντικά η ανεργία αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις χώρες εκείνες τις οποίες ε, ε, ο τομέας των κατασκευών είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία. Υπήρξε μια άμεση αντίδραση των χωρών, άμεση αντίδραση των χωρών μελών, των κεντρικών τραπεζών για να αποφευχθεί ε, η ε, αυτή ε, η τρομερή αναταραχή του οικονομικού συστήματος, ε, μια προσπάθεια λοιπόν προ την πραγματική οικονομία και αυτή η κρίση καταλαβαίνετε ότι είχε άμεση συνέπεια στα δημόσια οικονομικά. Μιλήσαμε για το... Πλέον δεν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά για το δημόσιο τομέα. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια κρίση και δημοσιονομική αστάθεια των δημοσίων λογαριασμών λόγω των ιδιαίτερων ξημένων ελλημάτων. Επίσης υπήρξε κρίση στο δημόσιο χρέος και αυτό βλέπουμε τους τελευταίους μήνες και όλα αυτά βέβαια επιδεινώνονται από δράσεις ε, ε, ε, των ιδιαίτερα ευάλωτων αγορών και μάλιστα από, ιδιαίτερα, από ιδιαίτερες κερδοσκοπικές επιθέσεις και όλα αυτά οδήγησαν σε σημαντική αύξηση Ε, του ε, ενδιαφέροντο των αγορών που στρέφουν τα βλέμματά τους προ τα κράτη, όταν τα κράτη προσπαθούν να πετύχουν ε, δανεισμό και αυτό έχει μετατραπεί πλέον σε πρόβλημα ολόκληρη Ευρωζώνη. Δεν είναι πλέον πρόβλημα ενός κράτους μέλους, αλλά αφορά τη σταθερότητα ολόκληρης Ευρωζώνη. Αυτά είναι τα γενικά πλαίσια. Ε, ε, ε, αυτά είναι με δύο λόγια τα γεγονότα και η διάγνωση που θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να δρά κατά συνέπεια. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά έδρασε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί να φάνηκε ότι υπήρξε μια βραδίτητα στη λήψη των αποφάσεων, απελπιστικά αργή όσον αφορά ορισμένες αποφάσεις, αλλά τελικά τα αποτελέσματα ήταν σωστά λογικά και χαρακτηρίζονται από μια σύνεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω συντονισμένη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που ε, τα επιμέρου μέτρα μα εμποδίζουν να δούμε το σύνολο, παρόλα αυτά νομίζω ότι ήταν σωστή η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των περιστάσεων. Ότι βεβαίω απαιτούνται κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα και ότι θα πρέπει ε, ταυτόχρονα να δούμε και το μεσοπρόθεσμα και το ε, μακροπρόθεσμο επίπεδο, αυτό είναι σίγουρο γιατί πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων κρίσεων ε, βραχυπρόθεσμα. Υπήρξε ε, μια ε, στάση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα σχέδιο συντονισμένο που έχει να κάνει με αυτή την άμεση δράση για να αντιμετωπίσουν τα άμεσα προβλήματα τα κράτη-μέλη και για να περιοριστεί, όχι για να εξαφανιστεί, να περιοριστεί το σύνολο ε, των ε, ζημιών που οφείλεται σε αυτήν την τεράστια κρίση. Μία εκδήλωση αυτή τη βραχυπρόθεσμη δράση σίγουρα είναι η βοήθεια προ την Ελλάδα, η περίπτωση τη Ελλάδα. Ήδη λοιπόν ε, πριν από μήνε είχε προειδοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε θα υπήρξε δυσκολία σε σχέση με τα δημόσια δημοσιονομικά τη χώρα αυτή. Και το Συμβούλιο απευθύνθηκε στην Ελλάδα με βάση το, το άρθρο 126.9 της Συνθήκης τη Λειτουργία τη ευρωπαϊκή Ένωση και προέβη σε μία σειρά συστάσεων και υποδείξεων και εξα... και ε, παρακολουθεί πολύ στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο την εξέλιξη των γεγονότων στην Ελλάδα. Ε, οι υποδείξει στην Ελλάδα δεν αφορούν μόνο τη ρευστότητα και τα δημόσια δημοσιονομικά, αλλά αφορούν ε, και μεταρρυθμίσεις, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, το συνταξιδοτικό σύστημα, ε, την ανάγκη να προβούν σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, την υγειονομική περίθαλψη και τελικά φτάνουμε στις 23 Απριλίου, εκεί όπου εγκρίθηκε ένας μηχανισμός παρέμβασης προς την Ελλάδα και μάλιστα αυτός ο μηχανισμός χθες οδήγησε σε μια πρώτη ε, σαφή ενέργεια με μια πρώτη αποστολή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αυτού του μηχανισμού ε, σωτηρίας, του συντονισμένου μηχανισμού προς την Ελλάδα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πρώτη έκφραση αυτή τη βραχυπρόθεσμη βοήθεια προ ένα κράτο μέλο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρέ δυσκολίε. Στη συνέχεια και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο πάλι ξεκινά και αυτό είναι μία από τις ε, εκδηλώσεις που εκφράζονται ε, σαφώς και που έχει να κάνει και με την ε, προφορική ερώτηση των Ντόλβε Χόσταντ ε, Σούλτς και άλλων προς την ανάγκη να υπάρξει μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Και η στρατηγική αυτή θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη, ε, ισόρροπη, που βεβαίως θα πρέπει να έχει ως στόχο την αποφυγή σοβαρών δυσκολιών ε, στα δημόσια δημοσιονομικά, αλλά ταυτόχρονα ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Αλλά κοιτάξτε, δεν αρκεί το βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όπω το είπαμε. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σε μέσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Διότι υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Προβλήματα τα οποία σε τελευταία ανάλυση αποδυναμώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη μια κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρών ε, οικονομικών αναταραχών. Και ε, θα, ε, ήδη λαμβάνονται μέτρα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, τα οποία είναι σημαντικά και θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Πρώτα απ' όλα διότι τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν να αποκριθούμε σε τέτοιε κρίσει όπω αυτή η σοβαρή οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση που, όπω είπαμε, αφορά το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω ε, αφορά ε, καθ' ολοκληρία την Ευρωζώνη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να, να ανταποκριθούμε ε, και να απαντήσουμε στην κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει, εφαρμόζει μία σειρά από μέτρα που συζητούνται ε, αυτέ τι ημέρε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα πακέτο εποπτεία, το οποίο πιστεύω ότι θα εγκριθεί ω το πιο γρήγορα και θα υπάρξει συμφωνία ε, μεταξύ των θεσμών, των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ένα μέτρο ε, το οποίο εγκρίθηκε και χτες από το ΕΚΟΦΗΝ. Η ρύθμιση δηλαδή των λεγόμενων hedge funds, των εναλλακτικών ε, κεφαλαίων, των κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Και εδώ αναφέρομαι και στην ερώτηση Hans Convedit που αναφέρονται ιδιαίτερα στο ζήτημα αυτό. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική ανάληψη δράσης στη G20, και εδώ ε, προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει να σα πω, είπαμε ότι υπάρχουν διαθετικέ αδυναμίε και ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ αυτό σκοπεύει η στρατηγική 2020-2020 που αφορά τη δέσμευση των κρατών μελών να ε, ασχοληθούν με συγκεκριμένου στόχου μέσα από μία σειρά ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών που θα ε, συνοδεύονται και από εθνικά προγράμματα ε, τα οποία θα ενσωματώνονται στα λεγόμενα ε, σχέδια μεταρρύθμισης. Και ταυτόχρονα είναι σημαντική η δράση του συνολικού ε, παραγωγικού συστήματος και εδώ σας παραπέμπω στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Μαΐου που μιλά για συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Η στρατηγική λοιπόν 2020 θέλει να ανταποκριθεί σε ένα ουσιαστικό ζήτημα το οποίο αφορά συνολικά το παραγωγικό σύστημα έτσι ώστε στο μέλλον να μην έχουμε τέτοιες αδυναμίες και να υπάρξει με περισσότερη ανταγωνιστικότητα ε, τη ε, οικονομία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωση, ε, φροντίζοντα και την προσθέμενη αξία μέσα από την τεχνολογία, κοινωνικές επιπτώσεις εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, απασχολησιμότητα και βεβαίω καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αφορά μόνο ε, τις παραγωγικές δομές του ιδιωτικού τομέα, αλλά αφορά και τα δημόσια οικονομικά. Και εδώ ε, θα σας αναφέρω άλλη πτυχή των μέσων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα δηλαδή τα οποία βρίσκονται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12 Μαΐου που χθε άρχισαν να συζητούνται στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, ε, στο Συμβούλιο λοιπόν των Υπουργών ε, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την εκπλήρωση των όρων του Συμφώνου ανάπτυξη και σταθερότητα, καθώ επίση ε, στα μέτρα επίλυση ή πρόληψη των κρίσεων. Με αυτή την έννοια ε, δημιουργήθηκε αυτή η Task Force, η οποία θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στι 21 Μαΐου, ε, την Παρασκευή, υπό την προεδρία ε, του ε, Προέδρου Βαν Ρομπάι και ακριβώ το βασικό θέμα θα είναι η δημοσιονομική πειθαρχία και η αξιοποίηση του εγγράφου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών ε, που έθεσε ο Επίτροπος Όλυ Ρεν. Αυτά τα μέτρα λοιπόν είναι περισσότερο μακροπρόθεσμου ε, χαρακτήρα. Και εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη συζήτηση των προβληματισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα για, ε, στο φορολογικό επίπεδο και κάτι το οποίο αρχίζει να συζητάτε ήδη ε, και σε επίπεδο G20 ε, και έχει να κάνει με τη φορολογία των ε, οικονομικών συναλλαγών και το οποίο ήδη συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο το ε, τονίζουν ιδιαίτερα και, ε, ε, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χάρμς και Κονβεντίτ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι όλοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή. Συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου ανατέθηκε μία μελέτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ε, τη φορολογία των ε, διεθνών αυτών ε, συναλλαγών. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο του Μαρτίου. Το έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Απριλίου και χθε επίση συζητήθηκε το ζήτημα αυτό στο Συμβούλιο Κοφίν. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε απέναντι σε ένα άλλο μέτρο το οποίο σίγουρα θα συστηθεί και σε επίπεδο G20. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέτρα ε, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Χθε, για παράδειγμα, στη συνεδρίαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Λατινική Αμερική, στη Μαδρίτη, ετέθη το σύστημα ε, τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Άρα το θέμα αυτό το θέτει σε όλα τα φόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή δημιουργούμε τις συνθήκες προς ε, την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συζήτηση αυτή συμμετέχει ιδιαίτερα ενεργά το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει ως ε, νομοθετικό όργανο και ως εποπτικό όργανο. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε με αυτά τα λόγια μου, ότι είναι αλήθεια ότι η κρίση τόνισε τις, και έδειξε τις ανεπάρκειες της Νομισματικής Ένωσης στην Ευρώπη. Προφανώς, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα οικονομική ένωση. Η οικονομική ένωση που προβλέπεται στις συνθήκες, αλλά δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Σταθήκαμε στην, σταματήσαμε στην Νομισματική Ένωση και δεν περάσαμε στην Οικονομική Ένωση. Τα βράχη πρόθεσμα αλλά και τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα σαφώς οδεύουν προς την κατεύθυνση της Οικονομικής Ένωσης. Πρόκειται για μια κρίση η οποία αποδυνάμωσε τις οικονομίες μας, η οποία ε, έθεσε ε, σε δοκιμασία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν την κατακαιρμάτισε και ε, δεν την αποδυνάμωσε. Ανταποκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με βραδύτητα αλλά με αξιοπιστία και ασφάλεια. Μερικές φορές φάνηκε ότι αμφιταλαντεύεται, αλλά πάντως προχώρησε ενωμένα. Και η απάντηση ήταν ορθή, ήταν λογική, ήταν σωστή, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της στιγμής. Και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να ε, σταθεροποιήσει αυτή την πορεία προς την οικονομική διακυβέρνηση, προς μια ενωμένη αντίδραση απέναντι στην κρίση ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα θα πρέπει να υπάρξει σωστή προετοιμασία τη κοινή θέση Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην συνεδρίαση των G20 στο Τορόντο για την ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και ε, όσον αφορά τη σοβαρή αυτή συζήτηση για την φορολογία των διεθνών οικονομικών συναλλαγών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την ε, παρουσίασή του εξ ονόματος ε, της, για την ε, Επιτροπή. Δίνω τον λόγο στον Επίτροπο Όλιρεν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, χαιρετίζω αυτή τη συζήτηση ε, για την ε, κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης. Θα αρχίσω ε, με τα άμεσα μέτρα και την απόκριση στην κρίση. Πριν από δέκα μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε θαραλέα μέτρα για την σταθερότητα στην Ευρώπη. Ήταν μια διτή απάντηση στην επιδεινούμενη κρίση η οποία είχε γίνει πρόκληση κατά του ευρώ. Επρόκειτο για μια αντίδραση που θα ονόμαζα σύμφωνο παγίωσης, δρέωσης, για έναν μηχανισμό σταθερότητας για εξυγίανση, το οποίο περιλαμβάνει 500 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που θα συμπληρωθεί με κονδύλια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεύτερον, συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε αυτά τα μέτρα εξυγίανσης στα κράτη-μέλη όπου τα μέτρα αυτά χρειάζονται περισσότερο και με κατεπήγοντα τρόπο. Η Ευρώπη κατέληξε σε ένα πακέτο αξιόπιστο που έδειξε στους πολίτες μας, στους αγορές και στον κόσμο ότι θα υπερασπιστούμε το ευρώ, το κοινό μας νόμισμα, με οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται. Δεν το κάνουμε αυτό για τις δυνάμεις της αγοράς, αλλά ε, για την αηφόρο ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας ε, ότι η σταθερότητα αυτή δεν θα ανακόψει την ανάκαμψη η οποία λαμβάνει η χώρα τώρα. Αυτή είναι η ευθύνη μας σε σχέση με τους πολίτες μας. Και με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο λαμβάνουμε μέτρα χτες ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ε, έχουμε, έχω, δώσαμε, εκταμιεύσαμε 14 δισεκατομμύρια, ευρώ για την ε, Ελλάδα και είπαμε ότι θα ήμασταν έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις άμεσες ανάγκες αναχρηματοδότησης της Ελλάδος και εκταμιεύσαμε εγκαίρως τα χρήματα αυτά. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται υπό όρους για με την εφαρμογή του προγράμματος που έχει σχεδιαστεί με την ελληνική κυβέρνηση ε, την ε, Επιτροπή, ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση του ευρώ. Εκτός από αυτά, τα κράτη-μέλη μας έχουν κατανοήσει την εξέχουσα σημασία αυτής της εξυγίανσης για να εξασφαλιστεί η αηφορία των δημοσίων οικονομικών που είναι προϋπόθεση ε, για την σταθερότητα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία παρουσίασαν ε, σημαντικά μέτρα ε, εξυγίανσης ε, οικονομικής και δημοσιονομικής που είναι δύσκολα μέτρα, σκληρά μέτρα, αλλά απαιτούμενα βήματα, απαραίτητα βήματα για να αντιμετωπιστούν αντιμετωπιστεί η εκτίναξη των ελλημάτων του 2010 και του 2011. Με την Επιτροπή θα γίνει μια αξιολόγηση της καταλληλότητας και της επάρκειας των μέτρων αυτών στις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα ήθελα να τονίσω ότι μια, συντο... μια ταχεία μείωση των ελλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το Σύμφωνο Σταθερότητος που συμφωνήθηκε στις 10 Μαΐου από το ΕΚΟΦΗΝ. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό οι δύο χώρες να υιοθετήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε ευξημένη οικονομική ε, μεγέθυνση ε, και θα μπορέσουν να εξηγιάνουν τα συνταξιοδοτικά και υγειονομικά συστήματα. Βεβαίω, είναι άμεση προτεραιότητα αυτή η οικονομική εξυγίανση στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συντονίσουμε τι οικονομικέ και δημοσιονομικέ μας πολιτικέ, ε, εφαρμόζοντα διαφοροποίηση ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν ε, τα μέτρα εξυγίανσης ανάλογα με τον, με τον ευάλωτο χαρακτήρα της οικονομίας. Οι χώρες οι οποίες έχουν λίγο δημοσιονομικό χώρο θα πρέπει να επιταχύνουν ε, τα μέτρα ενώ οι άλλες οι οποίες δεν έχουν ε, τέτοιο περιθώριο θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα ε, τα οποία χρειάζονται ε, για την, ε, την ενεργεία στην Ευρώπη. Θα ήταν λάθος να σταματήσουμε εδώ. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα πρώτα δέκα χρόνια του ευρώ ήταν μια ιστορία επιτυχίας. Αυτό είναι το σημείο κίνησης, αλλά η κρίση κατέδειξε ότι είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε τα, τις συστημικές ελλείψεις διότι τα μέτρα αυτά δεν μειώνουν το δημόσιο χρέος και αγνοούνται οι οικονομικές ανισορροπίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ε, στις 3 ε, Μαΐου η Κομισιό παρουσίασε ένα φιλόδοξο ε, φάσμα μέτρων για την Ευρώπη. Θέλουμε να ενισχύσουμε την προληπτική εποπτεία, την δημοσιονομική, να ασχοληθούμε με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και να θεσπίσουμε ένα μόνιμο στερεό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Επαφίεμαι ε, στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτές τις προτάσεις ούτως ώστε η Ευρώπη 2020 να γίνει επιτυχία στα επόμενα χρόνια. Οι προτάσεις μας βασίζονται σε δύο αρχές Πρώτα απ' όλα η πρόληψη είναι καλύτερη από τη διόρθωση για να ε, μην μιλήσουμε για το θέμα της κλιμάκωσης της κρίσης όπου είδαμε. Πρέπει να αποφευχθεί τέτοια κλιμάκωση. Η προληπτική λοιπόν εποπτεία και επιτήρηση πρέπει να συνοδεύεται με μακροοικονομική επιτήρηση ε, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί αηφόρος ανάπτυξη. Οι προτάσεις μας βασίζονται σε τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχύσουμε την προληπτική και διορθωτική αντιμετώπιση ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτή η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρέπει να συντονίσουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές ούτως ώστε οι εθνικοί προϋπολογισμοί ε, να είναι σύμφωνοι με και να συνάδουν με τις πολιτικές και υποχρεώσεις που υιοθετήσαμε, ούτω ώστε να μην κινδυνεύει η σταθερότητα της Ευρωζώνης στο σύνολό της και η σταθερότητα των άλλων κρατών μελών. Ας είμαστε σαφείς σχετικά με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ελέγχουμε ε, τους προϋπολογισμούς γραμμή προς γραμμή. Δεν έχουμε ε, πρόθεση ούτε πόρους προς το σκοπό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα αναλύουμε ε, και θα εξετάζουμε τις ευρείες κατευθυντήριες γραμμές και τις ισορροπίες ε, των προϋπολογισμών προτού να υποβάλλονται στα κοινοβούλια αυτοί οι προϋπολογισμοί με το νομικό δικαίωμα που βασίζεται στη συνθήκη να κάνουμε συστάσεις και να ζητούμε διορθωτικά μέτρα από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Μερικοί κατέκριναν αυτήν την πρόταση, ότι αυτή είναι παραβίαση δημοσιονομικής ε, ε, εθνικής κυριαρχίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω μπορεί να το κρίνει αυτή βεβαίως. Ε, έχουμε πλήρη συνείδηση της ευαισθησίας των εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα αυτό. Δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα ή την κοινοβουλευτική κυριαρχία, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη μας να μπορούν να σεβαστούν τους κανόνες τους οποίους προαποφάσισαν. Δηλαδή, να ε, το εφαρμόσουμε αυτό. Πρέπει να εισαγάγουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση στα οικονομικά. Δεν είναι ε, καλό να βλέπουμε μόνο εκ των υστέρων τι έχει γίνει με τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωζώνη. διότι οι εθνικές αποφάσεις έχουν επιπτώσεις πέραν των εθνικών ε, συνόρων, γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ε, συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από αυτές τις εθνικές αποφάσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι να προχωρήσουμε πέραν της δημοσιονομικής επιτήρησης ε, και να εξετάσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, γιατί αυτό είναι σημαντικό έχουμε ένα, μια διαφορά, ένα χάσμα ανάμεσα στις χώρες που είναι ελεματικές και στις χώρες που είναι πλεονασματικές και το χάσμα αυτό έχει διευρυνθεί ε, και αυτό βρίσκεται στην απαρχή της κρίσης ε, που ζούμε και που ζουν κυρίως μερικά από τα κράτη-μέλη μας. Πρέπει να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τα κατεπήγοντα προβλήματα προτού να εμφανιστούν και να κλιμακωθούν. Θα πρέπει να βρούμε δείκτες και τρόπους βαθμολόγησης και αξιολόγησης και να κάνουμε συστάσεις και να έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αν αυτό χρειάζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ε, ορισμένα μέτρα σχετικά με τις εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είναι προφανές ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ε, αποδυναμώσουμε την κατάσταση και κυρίως την εξαγωγική κατάσταση των χωρών θέλουμε να επανισορροπήσουμε τις, την, τα ισοζύγια αυτά στην Ευρώπη στο σύνολό της, πρέπει να ενισχύσουμε την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα όπου αυτό χρειάζεται και την εσωτερική ζήτηση όπου αυτό χρειάζεται και είναι εφικτό. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να παίξουμε ως Ευρωπαϊκή Ομάδα προ όφελος όλης της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι Όλος ο κόσμος παρακολουθεί ε, την Ευρωζώνη για να αποθαρρύνουμε τους άλλους να προσπαθήσουν να μας καταπολεμήσουν. Χρειαζόμαστε ένα, ένα πλαίσιο καταπολέμησης και διαχείρισης των κρίσεων για την Ευρωζώνη. Ο προσωρινός μηχανισμός της 10ης Μαΐου είναι ένα θαραλέο πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και μακροπρόθεσμα η Επιτροπή θα προτείνει έναν πιο μόνιμο μηχανισμό υπό ερεσιμότητα και αντλώντας τις διδάγματα από το πρόσφατο παρελθόν. Ναι, θα πρέπει να αποφύγουμε περισσότερους κινδύνους. Γι' αυτό ο μηχανισμός αυτός ε, θα πρέπει ε, να είναι χρήσιμος, αλλά η πρόσφατη ε, εμπειρία μας έδειξε ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα επίγουσης κατάσβεσης του πυρός για να μην το, η φωτιά γίνει πραγματικός κίνδυνος. Θα πρέπει να έχουμε μέτρα προστασίας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, για να εγκατακλείδει οι προτάσεις αυτές της Επιτροπής έχουν διανοίξει ε, τον ε, δρόμο ε, για την καλή οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε ένα σημαντικό σημείο, σημαντικό θέμα την ίδια μέρα που λάβαμε τις προτάσεις αυτές σχετικά με την αίτηση της Ιδεστονίας να γίνει μέλος της Ευρωζώνης. Ενώ το μέσο χρέος στην Ευρώπη είναι για την ώρα γύρω από το 75% ε, στην Εστονία όχι, είναι, δεν είναι 75, αλλά 7,5% σε διαρκή βάση. Αυτή η πρόταση ε, στέλνει ένα μήνυμα σημαντικό σε όλη την Ευρωζώνη ε, και μας δίνει εμπιστοσύνη και σκεφτόμαθα ότι θα μπορούν αυτές οι διαρκείς ε, πολιτικές ε, να αποφέρουν καρπούς. Οι προτάσεις ε, θα εμβαθύνουν στην οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και θα επιτρέψουν τη διεύρυνση της Ευρωζώνης. Στην ΟΝΕ είναι ήρθε ο καιρός να δώσουμε ζωή σε αυτό το οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τη δήλωση αυτή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ντόλ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτέλου η Ευρώπη αντέδρασε και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων άρχισαν αυτή τη στιγμή να κατανοούν το μέγεθο του προβλήματο και πριν από δέκα ημέρε αποφάσισαν ένα σχέδιο ε, σωτηρία του νομίσματό μα, του ευρώ. Ένα σχέδιο το οποίο μεταφράζει συγκεκριμένα την αλληλεγγύη ε, ει ε, πείσμα όλων όσων είχαν αμφιβολίε. Ένα σχέδιο όμω το οποίο δεν αρκεί και θα πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα μείωση των εθνικών δημοσιονομικών έλλειμμα από ε, μέτρα ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης ε, και συντονισμού σε επίπεδο 27 χωρών. Κοιτάξτε, εδώ και αρκετές ημέρες λέμε όλοι τα ίδια. Επιτέλους, ας τα εφαρμόσουμε. Σχέδιο το οποίο την περασμένη Τετάρτη συμπληρώθηκε από την απόφαση για να μειωθούν, για να ενισχυθεί δραστικά η εποπτεία και η ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητες. Κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση χωρί τα μέτρα αυτά. Ε, και απαιτείται ταυτόχρονα πολιτικό θάρρο. Διότι τα μέτρα τα οποία ήδη μπορέσαμε να λάβουμε συλλογικά και σε επίπεδο Ευρώπη αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ε, ε, τα, μέτρα τα οποία συζητάμε θα πρέπει να τα πάρουμε τώρα. Και αυτό αφορά όλε τι κυβερνήσει, και τι δεξιέ και τι αριστερέ. Θάρρο το οποίο δεν είχαν και πρέπει να το τονίσω και οι σοσιαλιστές της Γερμανίας όταν ψήφισαν το σχέδιο ε, θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να μάθουμε την αλήθεια ε, για, τις, για, τους για τα εθνικά δημοσιονομικά, όπως επίσης και για τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και, να, και όχι μόνο να καταγγέλει δειλά οποιοδήποτε κράτος μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά να το τιμωρεί. Κοιτάξτε, όλοι φοβόμαστε τα ραντάρ, όλοι φοβόμαστε τι κυρώσει, όλοι φοβόμαστε τους ε, πόντους που συσσωρεύονται στα διπλώματα οδήγησης. Θα πρέπει τώρα ε, όμως να αναλάβουμε σοβαρή πολιτική για την αντιμετώπιση όλων αυτών. Δεύτερον, οι 27 θα πρέπει να συντονίσουν τους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτησε την περασμένη εβδομάδα και εγώ ίδιος το ζήτησα ε, πριν από λίγες εβδομάδες στην αίθουσα αυτή. καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ε, εκνευρίζουν τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να Εμ. Ε, ε, να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση ε, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά τους σαν να ζουν το καθένα από μόνο τους σε ένα ερημικό νησί να μην καταλαβαίνουν ότι απαιτείται μια συντονισμένη δράση και αυτό βεβαίως ισχύει και σε επίπεδο κοινωνικών και φορολογικών πολιτικών γιατί μια άλλη μια φορά το λέω καταλαβαίνω το θυμό ορισμένων συμπατριωτών μας από τους οποίους ζητούμε να θυσιαστούν για τους υπόλοιπου που εργάζονται λιγότερο και που παίρνουν σύνταξη νωρίτερα και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί και αυτό είναι το τρίτο δίδαγμα το οποίο αντλώ από την κρίση αυτή. Το ευρώ θα είναι βιώσιμο μόνο αν όλοι φροντίσουμε γι' αυτό συλλογικά. Κοιτάξτε, ε, ε, εγώ δεν ζητώ ε, την, ε, τις οικονομικές συμβουλές του Προέδρου Ομπάμα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. τα εθνικά αντανακλαστικά θα πρέπει να αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά αντανακλαστικά. Οι κοντόφθαλμες πολιτικές που στοχεύουν στο να μην χάσουμε στις φυγμομετρήσεις σε εθνικό επίπεδο και να μην χάσουμε ψήφους θα πρέπει να μεταφραστούν σε άλλη νοοτροπία. Αυτό ζητούν και οι επενδυτές. Η ομάδα μου ζητά από την Ευρώπη να ξυπνήσει. Η ομάδα μου ζητά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει το καθήκον της. Δηλαδή ε, να εφαρμόσει τη θεραπεία στα κράτη-μέλη. Τη θεραπεία bonus μάλους όσοι, ε, να, να, να ανταμείβονται αυτοί που κάνουν το καθήκον τους και να τιμωρούνται οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει ότι υπηρετούμε τους Ευρωπαίους πολίτες και ότι υπηρετούμε τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα το οποίο τίθεται παντού αυτή τη στιγμή είναι το κατά πόσον ε, και αυτό που θέτουν οι πολίτες είναι το κατά πόσον ε, υπάρχει εγγύηση των καταθέσεών τους, των αποταμιεύσεών τους. Καταλαβαίνω τους πολίτες οι οποίοι εργάστηκαν όλη τη ζωή για να βάλουν λίγα χρήματα στην άκρη. Αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε πρώτα απ' όλα να του εγγυηθούμε. Το γεγονός ότι δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις τους, δεν κινδυνεύουν τα βιβλιάρια καταθέσεων. Και μόνο στα πλαίσια αυτά, κυρίε και κύριοι, η στρατηγική 2020 ε, θα έχει νόημα. Μόνο εάν ε, αποκτήσουμε σοβαρότητα, μόνο αν ε, αντιδράσουμε συλλογικά, θα κερδίσουμε τη μάχη κατά τη ανεργία, τη μάχη τη εκπαίδευση, τη κατάρτιση, τη έρευνα και τη καινοτομία. Το είπα χθε, το λέω κάθε μέρα. Εάν πρέπει να κάνουμε οικονομίε σε όλα τα κράτη-μέλη, τότε και εμεί οι Ευρωβουλευτέ και εμεί οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρέπει να δείξουμε το παράδειγμα, το καλό παράδειγμα. Διαφορετικά δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Αυτά έχω να σα πω. Κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει κρίσει ε, στο παρελθόν, βαθιέ κρίσει, σοβαρέ. Τουλάχιστον αυτή η κρίση να χρησιμεύσει για μια νέα αρχή για την Ευρώπη και για του πολίτε μα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα εξ ονόματος Τη σοσιαλιστική ομάδα, ο κύριο Σόλτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση σε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση τη διεξάγουμε. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που απειλείται σήμερα από αυτή την συγκυρία, από αυτή την κατάσταση. Δεκαετίες ολόκληρες είχαμε την ιδεολογία του laissez-faire στην Ευρώπη. Δεκαετίες όπου κάθε ένας όποιος θεωρούσε ότι είναι ανώτερο το καπιταλιστικό σύστημα, ότι αμφισβητούσε την ανωτερότητα του καπιταλιστικού συστήματος, εξοντωνόταν. Αυτό μας οδήγησε ως ιδεολογία στην πιο βαθιά οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση από τα τέλη του Δεύτερου Πολέμου και στην βαθύτερη ηθική κρίση και στην βαθύτερη κρίση νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τέλος του Δεύτερου Πολέμου. Αυτό το σύστημα είναι λάθος και είναι και όλας εν μέρη ανήθικο. Είναι στρεβλό. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για τι πράγμα κάνω λόγο. Διότι πολλοί από τους πολίτες μας δεν καταλαβαίνουν καθόλου την ορολογία που χρησιμοποιούν οι πραγματογνώμονες. Τι είναι το εμπόριο με CDS και τι είναι εκείνο το οποίο οδηγεί στην απώλεια ασφαλίσεων. Μπορεί να υπάρξει μια ασφάλιση που μπορεί κανείς να συνάψει ως αγαθό και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζει. Παράδειγμα, το ωραίο αγρόκτημα του κυρίου Ζωζεφ Ντόλ έχει μια ασφάλιση κατά αν τώρα αυτή την ασφάλιση, εγώ μπορώ να την, αυτό το συμβόλαιο κατά πυρός μπορώ να το αγοράσω εγώ, τον έχω στο χέρι και στην περίπτωση που καίγεται το σπίτι του πληρώνεται σε μένα ε, θα πληρωθεί η ασφάλιση και δεν χρειάζεται παρά κάποιος που να βάλει φωτιά στο αγρόκτημα του ντόλ και τότε θα έχω βγάλει λεφτά εγώ αυτό είναι ένα στρεβλό σύστημα και πρέπει να απαγορευτεί και να καταργηθεί όμως ε, Γι' αυτό το πράγμα, για αυτούς τους ε, μηχανισμούς ε, κάνουμε λόγο εδώ και συζητούμε. Και δεν είναι ευχάριστα παραδείγματα αυτά. Είναι ο τερματισμός των ε, συνταξιδοτικών ταμείων των ενώσεων διδασκάλων στην Καλιφόρνια διότι κάποιος ήθελε να αγοράσει μια αεροπορική εταιρεία. Δεν τα κατάφερε όμως κάτι άλλο αγόρασε. Το συνταξιδοτικό όμως αυτό το ταμείο των δασκάλων και καθηγητών ε, εξοντώθηκε και δεκαετίες που είχαν ε, συνεισφέρει καθηγητές και δάσκαλοι σε αυτό εξοντώθηκαν και διαγράφηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να ελεγχθεί σήμερα και να υπάρξουν πραγματικά μηχανισμοί ελέγχου. Τώρα καλούνται οι κυβερνήσεις να δράσουν με τα μέτρα που θα υιοθετήσουν. Ναι, το ακούσαμε από εσά κύριε Λόπε Γκαρίδο, το ακούσαμε από τον κύριο Ρεν. Όλα αυτά είναι ωραία λόγια. Μόνο όμω αντιδρούμε, αντιδρούμε. Είμαστε αγόμενοι και σειρώμενοι και φερόμενοι. Και αντιδρούμε πολύ με μεγάλη καθυστέρηση. Πολλά θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχουν γίνει και εμεί στην Ευρωβουλή το είχαμε ζητήσει. Έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί νωρίτερα. Τα hedge funds πρέπει να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Βαθμολόγηση, Αξιολόγηση. Είναι ομαλό όταν ακριβώς υπάρχει το ύψος της κερδοσκοπίας εις βάρος της Ελλάδας να υποβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας και να ακολουθεί η πιστοληπτική υποβάθμιση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να οδηγήσει σε κανόνες για αυτούς τους οίκους αξιολόγησης και πρέπει να ελεγχθούν. Έπρεπε πριν από χρόνια να έχουν γίνει αυτά. Εμείς το είχαμε απαιτήσει εδώ πριν από χρόνια. Απορρίφθηκε όμως. Είχε απορριφθεί από τις ίδιες κυβερνήσεις που σήμερα ζητούν ζητούν να είναι οι διαχειριστές στην οικονομική διακυβέρνηση αυτής της κρίσης. Διαμαρτυρίες εκτός μικροφώνου, δεν ακούγονται οι παρεμβάσεις. Κύριε συνάδελφε Λάγεν, ξέρω ότι σήμερα το απόγευμα θα καταθέσετε έτοιμα οι απόκριες να μην είναι ευκαιρία διεξαγωγής ολομέλειας στην Ευρωβουλή. Ωραίο αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν να συνεχίζετε με αυτού είδους παρεμβάσεις. Εδώ έχουμε διαρθρωτικά ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεσμικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε μια οικονομική νομισματική ένωση που δημιουργήσαμε, από ό,τι λέγεται. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δημιουργήσαμε μια νομισματική ένωση χωρίς οικονομική ένωση. Και έτσι υπάρχει μεγάλο κενό στην Ευρώπη. Στα 16 κυρίαρχα κράτη να μην έχουμε μια συντονισμένη οικονομική πολιτική και μάλιστα να είναι αντιφατική η πολιτική του ενός κράτους κατά του, άλλου κατά του άλλου αυτό είναι απαράδεκτο σε έναν ενιαίο νομισματικό χώρο. Μεγάλος κίνδυνος αυτός ο Σουάτσενέγκερ και η ε, Καλιφόρνια έχουν χαντακωθεί. Όμως ε, σε σχέση με, την, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό διακυβεύεται στην Ελλάδα, που δεν έχει αντιστοιχεία με τις ΗΠΑ, η κρίση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια οικονομική διακυβέρνηση. Όποιος είναι εναντίον δεν άκουσε τα σημεία των καιρών. Και έχουμε και μια κρίση πραγματικής νομιμότητας ε, και θεμητοποίησης. Ε, και οι πολίτες το ζουν αυτό. Βλέπουν ότι έχει αποτύχει το οικονομικό σύστημα και δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό. Και ζουν και βιώνουν ότι τα κρατικά θεσμικά όργανα που προχώρησαν αυτό το σύστημα και δημιούργησαν αυτή την κατάσταση είναι αγόμενα και φερόμενα και δεν έχουν πια εμπιστοσύνη σε αυτά τα θεσμικά όργανα πια. Σε αυτή τη φάση υπάρχει μεγάλος αριθμός που μία φυγή στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ζητούν μία διέξοδο στις ε, ρητορίες ε, των εθνικιστικών τόνων. Αυτές οι μεγάλες αντιφάσεις, ε, η απουσία εμπιστοσύνης στο οικονομικό μας σύστημα, στα θεσμικά κρατικά όργανα και η υποχώρηση, η παναχώρηση στα εθνικά θέματα πολλών θεσμικών οργάνων αντί να ζητηθούν οι λύσεις στα διεθνή θεσμικά όργανα και στις διεθνείς δομές, αυτό είναι κάτι το οποίο υπονομεύει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν για αυτούς τους λόγους μια οικονομική διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε επίσης ε, την δύναμη να περάσουμε και να υιοθετήσουμε τους δικούς μας κανόνες. Και τέλος, ο Ζωζεφ Ντόλ, όπου είναι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας ε, σε αυτή την κομματική ομάδα στο Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να ασκούν επικρίσεις εις βάρος άλλων. σας ευχαριστώ πολύ πολύ και τώρα εξ ονόματος της Συμμαχίας ε, <clears throat> των ε, Δημοκρατών ε, θα λάβει τον λόγο ο επόμενος αγορητής. Παρακαλώ κύριε Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι η ρητορική θα μας φέρει τις απαιτούμενες λύσεις για αυτή την κρίση. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μια νομισματική κρίση στην Ένωση, ούτε καν μια ε, κρίση του ενιαίου νομίσματος, αλλά μια κρίση της διακυβέρνησης της Ένωσης. Αυτό ζούμε σήμερα πρόκειται ότι θα έλεγα ότι είναι μια κρίση της εμμονής των κρατών μελών που νομίζουν ότι με, τους, με τη διακυβερνητική μέθοδο μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα στην Ευρώπη. Ενώ μια ζώνη νομισματική, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κυβερνάτε από μια ενιαία μέθοδο, να κυβερνάτε με τη μέθοδο την κοινοτική βάση του ευρωπαϊκού συμφέροντος και όχι από ένα συνδικάτο εθνικών συμφερόντων, το οποίο εκφύσεως είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ έχω τρία μηνύματα τα οποία θα ήθελα να εκφράσω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Γκαρίντο. πρώτα απ' όλα στο Συμβούλιο με το πρώτο μήνυμα και ζητώ από την Ισπανική ε, Προεδρία ε, να ζητήσει από τα μέλη να αρχίσουν να σωπαίνουν λίγο σε σχέση με την κρίση. Διότι κάθε φορά που βρίσκουμε μια λύση για να βοηθήσουμε το ευρώ, ο ένας ή άλλος αρχηγός κράτους ε, αρχίζει και δηλώνει ορισμένα πράγματα και αρχίζει να, να σαμποτάρει τη λύση που έχει βρεθεί. Ζητώ λοιπόν ίσως να σοπάστε λίγο στο Συμβούλιο, να αφήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βρεθούν λύσεις. Το δεύτερο μήνυμα που έχω το απευθύνω στην Επιτροπή. Νομίζω κύριε Ρεν ότι λάβατε αποφάσεις θαραλές την ε, περασμένη Τετάρτη προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η Επιτροπή. Για την ώρα έχουμε μια ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα συνεδριάσει ε, για να βρει λύσεις στο τέλος του Οκτωβρίου ή στο τέλος του χρόνου. Είναι πολύ αργά. Η Επιτροπή που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, έχει την υποχρέωση να υποβάλει ένα συνολικό πακέτο φιλόδοξο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα task force, μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εναπόκειται στην Επιτροπή να αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία για ένα πακέτο συνολικό που θα πρέπει να θέσει επιτάπητο για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο να ενισχύσει το Σύμφωνο Σταθερότητα. Χρειάζονται κυρώσει και εγώ νομίζω, ε, υποστηρίζω την ιδέα του κυρίου Ρεν και νομίζω και πολλοί άλλοι ότι στο πακέτο αυτό τα εθνικά κοινοβούλια, προτού τα εθνικά κοινοβούλια να εγκρίνουν ε, τον προϋπολογισμό τους, να υπάρξει μια παρακολούθηση, μια επιτήρηση, ένα σκρούτινι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι θέμα επικουρικότητας, αλλά είναι ε, θέμα πίστης, αφοσίασης στο ευρώ και στο σύμφωνο σταθερότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε μέλη του Συμφώνου και και της του ευρώ, αλλά ότι όσον αφορά τον προπολογισμό, εμεί δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε με το ευρώ. Ε, ότι είναι μια αρμοδιότητα καθαρά εθνική. Όχι, όχι. Νομίζω ότι στο πακέτο αυτό θα πρέπει επίσης να περιλάβουμε μια στρατηγική 2020 που να είναι πιστική. Και τώρα κύριε Γκαρίντο, ό,τι υπάρχει στο τραπέζι του Συμβουλίου δεν είναι πιστικό. Ε, θα καταλήξετε τον Ιωλά. Σε τι θα καταλήξετε. Θα καταλήξετε σε τι για τη στρατηγική 2020. Όπως με τη στρατηγική της Λισαβόνας που απέτυχε και πάλι. Έχουμε τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού. Αν είστε σοβαροί με το Συμβούλιο πρέπει τώρα να δώστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα μέσα, όλα τα όπλα, ούτω ώστε ε, να κατευθύνει η Επιτροπή την στρατηγική 2020, τη στρατηγική την οικονομική για να εξέλθουμε από την κρίση. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο που θα αντικαταστήσει ε, το μηχανισμό σταθερότητα που δημιουργήσαμε τώρα, διότι και εσεί, κύριε Ρέν το είπατε, αυτό ο μηχανισμό δεν θα επαρκέσει. Ο μηχανισμό αυτό είναι ένα μηχανισμό διακυβερνητικός χρειάζεται ομοφωνία για κάθε δανεισμό. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν κάθε τέτοια απόφαση. Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Τομείο που να το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επίτροπη και αναπαιτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι από τις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν κάθε φορά τα 16 κράτη-μέλη τους ε, Ευρωζών. Και χρειάζεται μια ομολογιακή αγορά ευρωπαϊκή αυτό περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται φιλοδοξία, θάρρο για να θέσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ένα πακέτο φιλόδοξο με αυτά τα τέσσερα ε, στοιχεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερη Συμμαχίας η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα εκ νέου αποφάσισε να υιοθετήσει μια θετική αντιμετώπιση, θετική στάση όσον αφορά τους μηχανισμούς ε, χρηματοοικονομικής ε, σταθεροποίησης που πριν από λίγο καιρό στις εβδομάδες ε, εγκρίθηκαν και συνδέουμε αυτή την υποστήριξη με μια σαφή ομολογία προς περισσότερες κοινοτικέ οικονομικές πολιτικές και περισσότερες κοινοτικές χρηματοπιστωτικές πολιτικές. Αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο για τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα. Ακολουθούμε μια πολυετή παράδοση από πλευράς μας. Συνδυάζουμε όμως αυτή την ομολογία πίστεως κύριε Ρεν Κύριε αξιότιμα εκπρόσωπε της Ισπανικής Προεδρίας, συνδέουμε αυτό το αίτημα με ένα άλλο αίτημα. Τώρα, επιτέλους, με σοβαρό τρόπο να αποφασίσουμε σε ευρωπαϊκό κοινοτικό επίπεδο να μην συνεχίσουμε μόνο να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα της κρίσης και να προσπαθούμε να τα θεραπεύσουμε, αλλά να αντιμετωπίσουμε την κρίση στις πλήρεις διαστάσεις της. Η ανάλυση μας δείχνει και λέει ότι από το 2008 ήδη είχαμε συμπτώματα τα οποία θεραπεύουμε. Από το 2008 και είχαμε χρεοκοπίες και τι κάναμε, θελήσαμε και σώσαμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και πρέπει να το πούμε αυτό και <clears throat> δεν σταθεροποιήθηκε πρόσφατα το ευρώ. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το προπροηγούμενο Σαββατοκύριακο, πάρα πολλές ε, τράπεζες γαλλικές και γερμανικές διασώθηκαν και στις ε, ισοτιμίες και στις συναλλαγές των χρηματιστηρίων είδαμε το τι συνέβη. Όμως από αυτή τη διάσωση πρέπει να εξέλθουμε πλέον, να βρούμε μια διέξοδο. Μας κοστίζει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων και δεν ξέρουμε από πού να αντλήσουμε αυτά τα δισεκατομμύρια πλέον. Και όταν την συμφωνία, για παράδειγμα, στο ΕΚΟΦΗΝ την δίκανης, τότε είναι μικρότατα, πολύ ελάχιστα βήματα <clears throat> όσον αφορά τις ε, ρυθμίσεις ε, στις ε, αγορές. Και τι βλέπουμε, αυτό, αυτό βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ετοιμάτων μας. Το κράτος πρέπει να επιστρέψει με στεναρότητα στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές αγορές. Δεν επιτρέπεται οι τράπεζες και οι κερδοσκόποι τους οποίους βρίζουμε εκείνοι να μας οδηγούν στο να γονατίζουμε εμείς μπροστά τους. Πρέπει αυτό το σύστημα το οποίο πάσχει σε βάθος να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση και να οδηγούμαστε επί ξηρού ακμής στα όρια της επιβίωσης. Ε, και θέλω να συνοψίσω. Για μας έχουμε κάποια πράγματα τα οποία σαφώς πρέπει να αποφασιστούν. Υπάρχουν μηνύματα ότι σε κάποια κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύουμε προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως ε, πρέπει να απαγορευτούν ε, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και hedge funds να ελεγχθούν επιτέλους τα κερδοσκοπικά κεφάλαια και να εισαχθεί ένα τέλος χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συναλλαγών. Δεν επιτρέπεται να εκφωνούμε δεκάρικους λόγους. Χρειαζόμαστε αυτό το τέλος επί των οικονομικών συναλλαγών, ώστε αυτά τα χρήματα τα οποία θα εισπραχθούν να μπορέσουν να αναχρηματοδοτήσουν δράσεις. Η συμμετοχή των κερδοσκόπων ε, θα, δεν επιτρέπεται να ε, συνεχιστεί. Πρέπει με την εισαγωγή αυτού του τέλους ε, χρηματοπιστωτικών αλλαγών, συναλλαγών να προχωρήσουμε στεναρά εναντίον τους και έτσι το μέλλον θα πρέπει να βρίσκεται υπό ένα συντονισμένο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την δημοσιονομική πειθαρχία. Ξέρουμε πολύ καλά αυτόν τον όρο, δημοσιονομική πειθαρχία από την Ομοσπονδιακή Γερμανία, στη, σε συνδυασμό με την ε, διαχείριση της κρίσης και μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής, της πολιτικής της Ευρώπης 2020 πρέπει να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε τι είναι αυτό που επιθυμούμε εμείς, πώς τα κράτη-μέλη, η Ευρώπη θα ανταποκριθούν στους πολίτες μας σε πέντε ή 10 χρόνια θα παρουσιαστούν ενώπιον των πολιτών στο επίπεδο της ευθύνης και υπευθυνότητας του κράτους. Η ευρωπαϊκή στρατηγική να είναι τώρα να ε, ακολουθήσουμε μία πορεία που θα οδηγήσει σε εξυλαστήρια θύματα. Τι θα γίνει με τα πανεπιστήμια, με τα παιδιά, με την ασφάλιση της συνταξιοδότησης των πολιτών, με τον πολιτισμό. Συνάδελφος Μπεντίτ είπε πρόσφατα ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμα εξυγίανσης. Εν τω μεταξύ γνωρίζουμε την ολέθρια οικονομική κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη πέρα από την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο για να δούμε πώς θα πορευθούμε στο μέλλον. Και όπως είπαμε, δεν θα πρέπει να περικοπούν οι κοινωνικές πολιτικές και να είναι η κοινωνική πολιτική το εξυλαστήριο θύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να είμαστε συνετοί στις, ε, στα δημοσιονομικά μας προγράμματα, να είμαστε δίκαιοι έναντι των μελλοντικών γενεών. Έχουμε ως πράσινοι πάντα τέτοια προγράμματα και αιτήματα τα οποία προ, προωθήσαμε στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Τελευταία παρατήρηση. Η πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές. Αυτή να θεωρείται ως κάτι επουσιώδες, όπως αυτό διαφαίνεται ότι θα γίνει. Αυτό θα ήταν το σενάριο του διαβόλου, ένα, διαβολ, ένα σατανικό σενάριο που θα οδηγούσε σε ολέθρια κατάσταση. Πρέπει να είμαστε φιλοπεριβαλλοντικοί σε σχέση με την παραγωγή μα. Να υπάρξει αναδιάρθρωση των δημόσιων μεταφορών. Δεν πρέπει να αγνοηθούν όλα αυτά. Πρέπει να διασφαλίσουμε τι θέσει ε, εργασία και απασχόληση με σωστή διοργάνωση, με αηφορία και φιλοπεριβαλλοντικά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε κονδύλια. Και κυρίε και κύριοι, είναι ταμπού να κάνει κανεί λόγο για νέου φόρου. Εγώ όμω σα ε, ομολογώ ότι είμαι πεισμένη σήμερα ότι από τη σημερινή κρίση δεν θα μπορέσουμε να βρούμε μια διέξοδο αν συνεχίζουμε να έχουμε ταμπού όσον αφορά για το ρόλο του κράτους και την ανάγκη ευφυών φόρων. Αν αυτό το ταμπού δεν το παραβιάσουμε τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ημίνιου. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ο κύριος Κερκόπ, παρακαλώ. Uh, Πρόεδρε, ε, κυρίε και κύριοι, δυστυχώ ε, είναι χαρακτηριστικό όσων υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιστεύουν ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι η περισσότερη ολοκλήρωση. Αυτή η προσέγγιση όμω χάνει την ουσία. Αυτό το οποίο λείπει από την Ευρώπη συχνά δεν είναι περαιτέρω μηχανισμοί για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, αλλά η πολιτική βούληση για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ήδη έχουν αναλυφθεί αλλά που δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Γι' αυτό πιστεύω ειλικρινά ότι η πρωτοβουλία για την Ευρώπη 2020, που σίγουρα είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί ε, η οικονομική κρίση που διανύει σήμερα η Ευρώπη δεν θα πρέπει να στηριχθεί στην ίδια βάση. Όσον αφορά την κρίση στην Ευρωζώνη, μα λέτε ότι για να αποφύγουμε τέτοιε κρίσει στο μέλλον ε, χρειαζόμαστε, ε, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητε για να ελέγχει του προπολογισμού που αποφασίζουν οι κυριαρχέ κυβερνήσει και για να επιβάλλονται κυρώσει. Μα κοιτάξτε, υποτίθεται ότι ήταν διαθέσιμα τα μέτρα αυτά, αλλά δεν γίνεται σωστά ο έλεγχο. Η έλλειψη οι αρμοδιότητες και ικανοτήτων αυτών που ασκούν τον έλεγχο σημαίνει ότι ε, ε, εκεί υπάρχει το πρόβλημα και οι κυρώσεις προβλέπονται απλά ε, στερούνται αξιοπιστίας και δεν πρόκειται με αυτά τα οποία προτείνεται τα πράγματα να καλυτερεύσουν. Τα, τα καινούργια μέτρα δηλαδή θα, ληφθούν υπόψη με περισσότερη σοβαρότητα και κάτι άλλο όσον αφορά την, την, την αντιμετώπιση, την αδειοδότηση σε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό έρχεται σε αντίθεση με, τις, με τη λογική της Τη οικονομική διακυβέρνηση που υποτίθεται ότι εφαρμόζουμε. Εάν, ε, και, και αυτοί που επιλέγουν να είναι στην Ευρωζώνη, αλλά και για την ευρύτερη οικονομία, ε, όλοι χρειαζόμαστε το ευρώ να είναι επιτυχημένο. Αλλά αυτό σημαίνει οι πολιτικέ που εφαρμόζονται να είναι αξιόπιστε ε, και να εκπληρώνονται οι συμφωνημένε δεσμεύσει. Η Επιτροπή παραδέχεται η ίδια ότι οι προτάσει τη τώρα θα οδηγήσουν σε περισσότερη εμβάθυνση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση ε, όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφή του Μαρτίου. Το αγγλικό κείμενο αναφερόταν σε governance, σε διακυβέρνηση, ε, στο οποίο αναφέρεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά το γαλλικό ε, κείμενο αναφέρεται στη λέξη government, κυβέρνηση. Φαίνεται λοιπόν ότι η φιλοδοξία τελικά είναι αυτή. Με αυτόν τον τρόπο όμω δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ε, και θα δράσουμε ει βάρο των κρατών μελών, των πολιτών αλλά και τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Και τώρα, ε, εξ ονόματο τη ε, ενωτική Αριστεράς, ε, να δώσουμε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, οι τελευταίες σύνοδοι του Συμβουλίου δείχνουν ριζοσπαστικέ αλλαγέ. Αυτά τα οποία ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία κυβερνοποίησης ε, της ε, πολιτικής στην Ευρώπη. Στη Λισαβόνα όμως δεν αποφασίστηκε και επενέθηκε ο ρόλος και ενίσχυση της Ευρωβουλής και εμείς τον είχαμε επενέσει. Τώρα γίνονται σοβαρές ε, αλλαγές και συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων και τεράστια ποσά δαπανώνται τα κοινοβούλια μέχρι σήμερα δεν είχαν λόγο να αρθρώσουν επ' αυτής της διαδικασίας και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την, σε αυτή την τάση. Η μέθοδος που εφαρμόζουν οι κυβερνώντες είναι τεράστια κονδύλια για την διάσωση των ε, υπεύθυνων χρεοκοπημένων τραπεζών που οδήγησαν σε ένα καπιταλισμό καζίνου και τώρα διασώζονται. Η κρατική ε, αυτή διάσωση σε άλλους τομείς έχει καθυστερήσει. 750 δις ευρώ κάπου βρέθηκαν ξαφνικά. Το θέμα είναι ότι θα, θα τυπώνουν χρήμα. Ποιοι θα διασωθούν, τα κεφάλαια των τραπεζών πιστεύω πρώτα. Η Ευρωπαϊκή όμω Ένωση πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μια ελεύθερη ενιαία εσωτερική αγορά με ένα ενιαίο νόμισμα. Ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δίκιο όταν λέει χωρί μια ε, οικονομική ένωση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η νομισματική ένωση. Όμως δεν βλέπω κάποιο ξεκάθαρο πρόσωπο και ξεκάθαρες γραμμές όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ένα σοβαρό συντονισμό στα οικονομικά θέματα. Εδώ λείπει μια κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που απουσιάζει είναι η αηφορία και η ρύθμιση με στεναρό τρόπο του οικονομικού τομέα. Λείπει η φορολογική πολιτική και ο συντονισμένος ε, ε, ρόλος ε, της ανταμοιβή των εργαζομένων με σωστούς δίκαιους μισθούς. Ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή τα κοινωνικά θέματα να διασφαλιστούν από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να περικοπεί η πολιτική για τα κοινωνικά θέματα. Υπάρχει φόβος όσον αφορά και την Ελλάδα και άλλες χώρες όταν βλέπουν τις κοινωνικές περικοπές. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή να υπάρξει προσπάθεια εναρμονισμού σε υψηλά επίπεδα των κοινωνικών παροχών και των μισθών. Οι φορολογικές οάσεις πρέπει να καταργηθούν. Στην καταπολέμηση της οικονομικής χρηματοπιστωτικής κρίσης υιοθετούμε ρυθμούς χελώνας και με τις ταχύτατες κινήσεις των κερδοσκόπων αυτό δεν επαρκεί. Είναι μεγάλο σφάλμα στη σημερινή κατάσταση τα δισεκατομμύρια των απολειών να κοινωνικοποιούνται και τα κέρδη να είναι κέρδη ιδιωτικά. Δεν είναι δυνατόν άμεσα οι ε, φορολογούμενοι να πληρώνουν τα σπασμένα για την αποτυχία των τραπεζών. Και σήμερα με τις ε, σημερινές έννοιες ε, ο όρος ληστής, ληστής τραπεζίτης πρέπει να επανακαθοριστεί. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος των Δημοκρατών θα λάβει τον λόγο η κυρία Τζαβέλα παρακαλώ. Επίτροπε, δράτω με τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την σκληρή και αποτελεσματική δουλειά που έχετε καταβάλει για την οικονομική κρίση στην πατρίδα μου την Ελλάδα. Εξίσου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου για τη στήριξή τους και την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, έχω τρει προτάσει και θα ήθελα, κύριε συνάδελφοι, πολύ εμφαντικά να ζητήσω τη στήριξη των προτάσεων αυτών. όσον αφορά για την υιοθέτηση ενός μονίμου εργαλείου για την οικονομική διακυβέρνηση το ινστιτούτο Μπρούγκελ, το οποίο είναι ένα think tank επί οικονομικών θεμάτων προτείνει το εξής η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να εγγυάται ευρωπαϊκά ομόλογα ύψους μέχρι το 60% του ΑΕΠ κάθε χώρας. Τα ονομάζει blue bonds. Όσες υπερβαίνουν το 60% να δανείζονται με όρους αγορών για το ποσοστό της υπέρβασής τους, τα λεγόμενα red bonds. Αυτή είναι μια πρόταση για ένα μόνιμο εργαλείο στην οικονομική διακυβέρνηση δεν χρειάζεται να στήσουμε καινούριου μηχανισμούς κτλ. πολύ γρήγορα μπορεί να υιοθετηθεί. δύο ad hoc προτάσεις για την ελλάδα το διεθνές νομισματικό ταμείο θα παρατείνει την περίοδο αποπληρωμής του δανείου προς την ελλάδα από τρία έως πέντε χρόνια αν η ίδια παράταση χρόνου υιοθετηθεί ε, από τους ευρωπαίους δανειστές μας θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα και πιο ρεαλιστικά η ελλάδα να αποπληρώσει το χρέος της και αυτό θα είναι ένα καλό μήνυμα για τις αγορές. η δεύτερη πρόταση το ποσό της βοήθειας προς την ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή των ομολόγων μας. μια ορθολογική διαχείριση του θέματος θα ήταν η ευρώπη να απελευθερώσει από τώρα πόρους που μελλοντικά θα δώσει στην ελλάδα για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση αμήνεται μαζεύει λεφτά προσπαθεί να μαζέψει λεφτά για να μπορέσει να μειώσει το χρέος της. δεν έχουμε παράλληλη αναπτυξιακή προσπάθεια. γι' αυτό κύριε επίτροπε θα έλεγα αν μπορούσε να στηριχθεί και μια παράλληλη αναπτυξιακή προσπάθεια θα ήταν πολύ καλό. κλείνοντας κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να πω ότι ας ελπίσουμε η ελληνική κρίση να είναι το μόνο αντίτιμο που έχει να πληρώσει η ευρωπαϊκή ένωση για την επιτροχάδη ε, σύσταση της οικονομικής διαχείρισης που έπρεπε να έχει ε, τη οικονομική ε, κυβέρνηση που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και δέκα χρόνια. Α ευχηθούμε να είναι μόνο η ελληνική κρίση το τίμημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν σα διέκοψα επειδή είστε από την Ελλάδα, αλλά ήταν πάνω από ένα λεπτό περισσότερο από τον χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Δεν ήθελα να σας ε, διακόψω επειδή είσαστε από την Ελλάδα και μιλήσετε τόσο πολύ ε, για την Ελλάδα, αλλά την επόμενη φορά θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, όταν γίνατε πρόεδρος πέρσι αυτού του Κοινοβουλίου είπατε ότι θα αντιμετωπίζετε όλες τις ομάδες και τα κόμματα ε, με τον ίδιο τρόπο. Ο κύριος Σούλτς είχε 10 λεπτά περισσότερο. Ε, γιατί λοιπόν υπάρχει, υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις εναντίον μιας πολιτικής ομάδας. Θα ήθελα, ε, να σας πω το εξής. Όσον αφορά το χρόνο αγόρευσης, είναι αλήθεια ότι ορισμένοι μιλούν περισσότερο και μίλησαν περισσότερο. Αλλά εγώ τώρα αναφέρθηκα στην κυρία η οποία μίλησε πριν από ένα λεπτό, στην κυρία Τζαβέλα, η οποία ε, μίλησε πολύ περισσότερο. Ε, σεβάστηκα όμως το γεγονός ότι ε, είναι Ελίδα και σκέφτηκα ότι είναι σημαντικό να ε, μιλήσει λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο αγόρευση, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε βεβαίω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βάγνερ εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, ε έπρεπε να φτάσουμε στην άβυσο και στην οικονομική κρίση έτσι ώστε οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων να καταλάβουν ότι ε, ο δρόμο ε, που θα πρέπει να ακολουθήσουμε δεν είναι περισσότερο εθνικισμό αλλά περισσότερη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ε, κυκλοφορούν μέτρα ε, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με το βέτο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με αγορά ομολόγων στην Ευρώπη κτλ. Τέλο πάντων τελικά καταλάβαμε ότι όλοι στο ίδιο πλοίο βρισκόμαστε και ότι είναι ανώφελο να αντιμετωπίζουμε ευκαιριακά τις καταστάσεις και αυτοσχεδιάζοντας. Αυτοσχεδιάζοντας. Αναρωτιέμαι όμως, αυτή η στάση τι είναι, ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή ή απαρχή μιας πραγματικής ε, οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Γιατί, ε, κοιτάξτε, ε, ε, ε, ε, κυβέρνηση θα έλεγα. Διακυβέρνηση έχουμε παραπάνω από όσοι χρειαζόμαστε. Κυβέρνηση χρειαζόμαστε. Αυτό ήθελαν και οι πατέρε τη Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε όλε εκείνε τι μεταρρυθμίσει που στοχεύουν στο να ενισχύσουν την Ευρώπη και να την κάνουν σε μια πραγματικότητα και σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε επίπεδο δημοσιονομική πειθαρχία. Και α ξεχάσουμε τι νοσταλγίε ε, περί κυριαρχία, περί εθνική κυριαρχία. Κυρίε και κύριοι, ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο μόνο σωστό δρόμο για να οικοδομήσουμε με μία Ευρώπη. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα εξαλειφθεί, θα εξαφανιστεί ε, η Ευρώπη. Δεν θα υπάρχει πλέον. Θα σε ευχαριστούμε πολύ και τώρα άλλοι αγορητές θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι διεξάγουμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που θα επηρεάσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα λάβει τον λόγο κυρία Βόρτμαν Κόλ. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι εάν ε, το αγρόκτημα του κυρίου Ντόλ πιάσει φωτιά, πρέπει πρώτα απ' όλα να σβήσει τη φωτιά. Γι' αυτό η ομάδα μας συμφώνησε με τις προτάσεις ε, του Συμβουλίου. Λήφθηκαν αποφάσεις για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για ένα τέτοιο πακέτο. Αυτό ήταν αναπόφευκτο και μια εβδομάδα νωρίτερα έγινε λόγος για τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τους κανόνες τους δημοσιονομικούς. Το Συμβούλιο ήταν ομόφωνο, ας είμαστε και εμείς ομόφωνοι, αλλά όταν ακούω τον συνάδελφο κ. Σούλτ από την σοσιαλιστική ομάδα βλέπω ότι δεν έχουμε εδώ αυτή την ομοφωνία. Εμείς όλοι θέλουμε μια Ευρώπη με μια ανάπτυξη αηφόρο, διατηρήσιμη, με αρκετές θέσεις εργασίας για τους πολίτες μας, με υγιείς επιχειρήσεις. Αυτό θα καταστεί δυνατόν μόνο με ένα νόμισμα σταθερό και μια οικονομία σταθερή. Ε, για να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη στρατηγική 2020, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να γίνει σεβαστό. Αυτό είναι ένα κρίσιμο, ζωτικό θέμα και για να το κατορθώσουμε χρειάζεται μια στιβαρή οικονομική διακυβέρνηση και είναι το νόημα του ψηφίσματος που ετοιμάσαμε ε, με, τους, ε, με τις πολιτικές ομάδες. Θέλουμε να σας υποστηρίξουμε κύριε Ρέν και θα ήταν ανεύθυνο οι, οι συνάδελφοί μας, οι σοσιαλιστές, να μην δώσουν την υποστήριξή τους αυτές τις προτάσεις. Κύριε Πρόεδρε, Υπάρχει η ανεύθυνη στάση των κερδοσκόπων. Δεν είναι η αιτία όλων των προβλημάτων, αλλά αυτό επιδίνωσε την κρίση. Ο κύριος Μπαρνιέ πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά του, πρέπει να κάνει προτάσεις σχετικά με τις ανεύθυνες συμπεριφορές στις οικονομικες αγορές. Πρέπει να τεθούν όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χανές Βόμποντα παρακαλώ στη συνέχεια. Κύριε Σβόμποντα παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Βόρτμαν Κολ κάνει λάθος, διτό λάθος. Πρώτον, δεν θέλουμε να καεί το αγρόκτημα του κυρίου Ντόλ. Δεν θέλουμε κανένα αγρόκτημα να καεί. Θέλουμε προληπτικά να δράσουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Και δεύτερον, υποστηρίζουμε απόλυτα τα μέτρα τα οποία πρότεινε ο κύριος Στραέν μόνο που δεν, δεν επακούν. Και υπό αυτό το πρίσμα, μια και τα περισσότερα μέτρα τα οποία προτείνονται και προτάθηκαν έχουν οδηγήσει εντωμεταξύ στο να καίγεται το αγρόκτημα του κυρίου Ντόλ και είπαμε ότι πρέπει να παρακολύσουμε, να παρεμποδίσουμε το να καεί. Αυτός είναι ο στόχος. Και τώρα πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αργός ο ρυθμός λήψης αποφάσεων. Και έτσι η υπερβολική βραδύτητα οδήγησε στο να αντιληφθούν κάποιοι το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Ρεν σωστά ανέφερε ότι οι διαφορές που έχουμε στον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών μας ε, οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη παρέκκληση και όχι σε σύγκληση. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό το οποίο δεν αναφέρεται κύριε Ρέν και είναι πολύ σημαντικό είναι οι διαφορές μεταξύ φτωχών και πλουσίων στην Ευρώπη που αυξήθηκαν και όταν αυτό ακούγεται με αυτόν τον τρόπο για μας είναι ένα θέμα κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής πολιτικής. Κάποιους όμως δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα θέλουν οικονομικά μέτρα, αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία προτείνονται και έτσι οι άνθρωποι πιέζονται, οι πολίτες ε, βλέπουν ότι υπάρχει ανάπτυξη και διαφορά μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Αυτό δεν είναι ε, σωστό και δεν είναι δίκαιο και αποδεκτό. Γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες ε, και διαδηλώσεις. Πρέπει να βρούμε τα σωστά ισόρροπα μέτρα και γι' αυτό έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πρώτον, πρέπει σίγουρα τις διαφορές των ανταγωνισμών να τις μειώσουμε πάλι. Πρέπει να πετύχουμε και να το καταφέρουμε και έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Η ανταγωνιστικότητα χωρών όπως της Ελλάδας, της Ισπανία, τη Πορτογαλία πρέπει να αυξηθεί. Δεν θέλουμε εδώ να επιδεινωθούν και να γίνουν χειρότερε οι συνθήκε ε, ανταγωνισμού τη Γερμανία και άλλων χωρών. Αλλά βελτίωση των ανταγωνιστικών όρων και προποθέσεων. Αυτή είναι απόλυτα αναγκαία και σωστή στρατηγική. Μόνο που στην επικοινωνία σα και ανακοίνωση, κύριε Ρεν, λείπει εδώ, λείπουν συγκεκριμένα μέτρα. Πώ θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Και αναφέρατε μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία ε, και των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αληθέ δουλεύει αυτό, αλλά δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί να αναθεωρήσουμε την αγορά εργασία και τα συνταξιοδοτικά ε, συστήματα. Δεν επαρκούν. Αν δεν ε, αναδιαρθρώσουμε, δεν χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέτρα και μέσα στρατηγική ε, για την Ευρώπη του 2020, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και σα παρακαλώ αυτά τα δύο πράγματα να τα προσέξετε. Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική ασφάλεια. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ και στη συνέχεια η κυρία Βαλάν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη αλλά που εξακολουθούν ε, να συμμερίζονται τις ανησυχίες με τους υπόλοιπους. Οι πολιτικοί ηγέτες ε, στη χώρα μας αναφέρουν την ιδέα ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να αποτελεί ένα όπλο για την αντιμετώπιση των δύσκολων καιρών. Και όμως αυτή τη στιγμή το ευρώ αντιμετωπίζει επιθέσεις από όλες τις μεριές παρόλε τι προσπάθειες που καταβάλλονται. και κοιτάξτε, η εξαιρέσεις χρημάτων ε, αποτελούν μια ε, συγκυριακή αντιμετώπιση. Ας το αντιμετωπίσουμε, ας αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Το θέμα ε, είναι ότι δεν μπορούμε να διαφύγουμε από τη βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, διότι η έλλειψη ισορροπίας οδηγεί σε αυτές τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Για να υπάρξει λοιπόν η δημοσιονομική πειθαρχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούνται μηχανισμοί διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και ελέγχου. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, να προσελκύσουμε κεφάλαια, να μειώσουμε με θάρρος τις γραφειοκρατικές δαπάνες. Χρειαζόμαστε ε, αποφασιστικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Στη Ρουμανία για παράδειγμα η κυβέρνηση μειώνει τις συντάξεις ε, και του μισθού αντί να ε, μειώνει τα χρήματα τα οποία δαπανώνται, σπαταλώνται για ε, ψηφοθερικού σκοπούς κτλ. Ε, έχουμε συστήματα τα οποία είναι παρόμοια συστήματα της FBI και όμως ε, δεν μειώνουμε εκεί τι δαπάνε, αλλά τις μειώνουμε από τα σχολεία και από τα νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα και να, και, και να μην ξεχνάμε ότι μόνο λίγα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν το παράδειγμα σήμερα. Ευχαριστώ κύριο Λαμπέρ, ένα μισή λεπτό. Ναι, ε, κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, Χρειαζόμαστε υπεύθυνε δημόσιε δαπάνε. Πρέπει να εξισορροπήσουμε του προπολογισμού μα και χρειάζεται διαχείριση ε, υπεύθυνη των οικονομικών. Ενίσχυση βεβαίω αμοιβαία, αλλά όχι ε, κύριε του Συμβουλίου, κύριοι κυρίω και όχι τόσο κυρίε, αλλά είναι πλάνη ε, να αφήνουμε του άλλου να πιστεύουν ότι μόνο μειώνοντα τι δαπάνε θα ανταποκριθούμε στι προκλήσει, διότι αυτό θα οδηγεί στην Ευρώπη στην ύφεση ε, και θα καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό, την κοινωνική συνοχή που είναι μέρος της ε, ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αν θέλουμε να εξισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά δεν υπάρχει άλλη λύση και να μπορούμε και να επενδύσουμε διότι δεν πρόκειται μόνο για την μείωση των ελλημάτων πρέπει να επενδύσουμε στον μέλλον μας ε, και να βρούμε νέα έσοδα. Δηλαδή ο χρηματοπιστωτικός τομέας να συμβάλλει, φόροι στις συναλλαγές και θα πρέπει όσοι έχουν επωφεληθεί περισσότερο από, κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, από τα έσοδα, να πάψουμε να κάνουμε δώρα ε, σε αυτούς ε, τους πιο πλούσιους της κοινωνίας, στις επιχειρήσεις ε, οι οποίες έχουν ορισμένα πλέον εκτήματα φορολογικά και επωφελούνται. Και θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με ένα άλλο ταμπού, όχι το ταμπού το φορολογικό, αλλά της κυριαρχίας, το οποίο εσείς κύριοι και κυρίες του Συμβουλίου με την υποστήριξη ε, του ΕΛΚ υποστηρίζεται. Η φορολογική, την δημοσιονομική ε, κυριαρχία θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με τις αιτίε του προβλήματος. Θα ήθελα να... Ιωγιάν Έπινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Βεβαίω υπάρχει. Ονομάζεται φορολογικό συντηρητισμό. Το διορθωτικό τομείο, το πρόβλημά μα είναι ότι ε, οι δαπάνε του δημοσίου διέρχεσαν για πάρα πολύ καιρό και τα πράγματα έφυγαν από τον έλεγχο για πολλά χρόνια. Ε, η γερμανική κυβέρνηση του κυρίου Σρέντερ ε, είχε αναφέρει το, την οροφή του 3% και την ξεπέρασε. Και βεβαίω το ρεκόρ το κατέριψε η Ελλάδα. Γιατί δεν μπόρεσε να γίνει σωστή διαχείριση των χρημάτων. Συνέχεια είχαμε το Σύμφωνο Σταθερότητα. Τι είπε ο κύριο Πρόντι το 2002 για το Σύμφωνο Σταθερότητα. Το ξέρετε. Ε, ήσασταν στην κυβέρνησή σα τότε. Είπε ότι ήταν ανόητο. Άρα έπρεπε να το αλλάξουμε. Ε, αυτό το είπαν οι θεματοφύλακε τη συνθήκη. Το, το αλλάξατε. Και είδαμε τα αποτελέσματα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, πρέπει, ε, ε, πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του φορολογικού συντηρητισμού. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε καινοτομία, περισσότερε ελεύθερε αγορέ, περισσότερε δεξιότητε των επιχειρηματιών, κύριε Σούλτ. Χρειαζόμαστε φορολογία. Απευθύνομαι στην, στον πρόσωπο τη Ισπανία. Όχι, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε στασιμότητα. Και θα έχουμε το Ρομπέντο Δασόν από την ανάποδη, θα έλεγα. Άρα λοιπόν Καταλαβαίνω το θυμό των πολιτών, των συνταξιούχων, ε, των ανθρώπων που έχουν αποταμιεύσει. Καταλαβαίνω του Γερμανού φορολογούμενου. Ξέρουν ότι πρέπει να πληρώσουν. Αλλά οι Γερμανοί φορολογούμενοι δεν μπορεί να πληρώνουν ε, για πάντα. Και κοιτάξτε κύριε Βερχόστα, δεν ξέρω αν είστε ακόμα στην αίθουσα. Ε, δε, ε, ε τι να πείτε στην κυρία Μέρκελ να σταματήσει να μιλά για το ευρώ. Μα κοιτάξτε, πώς, ε, τι προσπαθεί να αποδείξει ο κύριο Βερχόφσταφ με αυτή τη στάση. Ο συνάδελφος Πατρίκλου Γιαρίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να καθησυχάσετε τις χρηματοπιστωτικές αγορές αν δεν ξαναγυρίσετε στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεμφαλαίων και του ελεύθερου ανταγωνισμού που είναι ανισότητα ανταγωνισμού. Σήμερα βάζουμε πολλά χρήματα πάνω στο τραπέζι αλλά για να καθυσυχάσουμε τις αγορές ενώ στους λαούς υπόσχεστε αίμα και δάκρυα. Ε, βάλατε το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στο στάβλο των Ευρωπαϊκών. Γιατί εμεί δεν μα συμβουλεύτηκαν για αυτήν την απόφαση και τώρα ε, θέλετε ένα πραγματικό σφετερισμό των εξουσιών ελέγχοντα ε, από την ίδια την Επιτροπή του εθνικού προπολογισμού, Μιλάτε για τα ελλείμματα και για τα χρέη συνεχώ. αλλά γιατί ποτέ δεν μα μιλάνε για την δυνατότητα των εσόδων που υπάρχουν. Διότι αν σήμερα υπάρχουν ελλείμματα είναι επειδή μειώνουμε συνεχώ την φορολογία του κεφαλαίου και δημιουργήσαμε τις συνθήκες μιας όλο και πιο άνησης κατανομής του πλούτου στα μέτρα που πρέπει να λάβουμε πρέπει να ε, τροποποιήσουμε το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χρειάζεται μια πραγματική αλληλεγγύη. Ο συνάδελφος Μάριο Μποργέζιο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο θα κρατήσει το ευρώ έτσι με τη σημερινή του μορφή μέσα σε ένα-δύο χρόνια ε, θα το αποδομήσουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι ε, αυτή τη στιγμή ε, ε με αυτά τα, τα συμπληρωματικά κονδύλια θα καλύψουμε τα πράγματα και, και δεν πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα αρκούν για να οικοδομήσουμε το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ με το δόγμα να σώσουμε το ευρώ με τη σημερινή του μορφή. Γιατί κοιτάξτε, ε, ε, εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ευρώ, με τα επιτόκια και το πώς θα διοχετεύσουμε ε, τα κεφάλαια προς τις επενδύσεις, προς τις βιομηχανίες μας, οι οποίες ασθμένουν αυτή τη στιγμή. και δεν συμφωνώ με το να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα, εξετάζει προληπτικά και, θα, και θα ελέγχει τους, προ, προπολογισμού πριν από τα εθνικά κοινοβούλια. Δηλαδή, αποχαιρετάμε τελείω την εθνική κυριαρχία στοιχεία. Δεν συμφωνώ με την οικονομική και την νομισματική αυτή ε, πολιτική. Διακόπτει ο πρόεδρο. Ε, Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ο Χάν Πέτερ Μάρτιν, παρακαλώ, στη συνέχεια. Θα ήθελα να στραφώ κατά της απαράδεκτης ε, Εχθρική ε, στάσης κατά της Ευρώπης του Συμβουλίου. Παραπονείστε για αυτή την κρίση και τώρα δημιουργείται οικονομικά προτεκτοράτα. Και όμως ε, είσαστε συνυπεύθυνοι για πολλά πράγματα. Δεν επιτρέψατε τι ρυθμίσει όταν ήταν αναγκαίε Για να δώσω ένα παράδειγμα, Ευρωστάτ, Eurostat και όσον αφορά επικρίσεις ε, που είχαν ασκηθεί έγκαιρα είχαν αναφέρει τα προβλήματα στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να ε, δημιουργηθούν ε, οι αναγκαίες ε, δράσεις έρευνας και τροχοπεδήθηκαν εσείς από την Ισπανία και σε σχέση με την Γερμανία και με την Γαλλία και μάλιστα και οι Αυστριακοί δεν ήθελαν να, να τους δουν να εξετάσουν τα βιβλία τους, τα λογιστικά βιβλία τους διότι ήξεραν ότι είχαν πολλά λάθη και ότι πολλά ε, είχαν χρεωθεί και κατά τα άλλα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ποινικέ ε, ε, κατηγορίες που έχουν εγερθεί όσον αφορά και την ίδια την κατάσταση στην Αυστρία. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε όμως ε, δεν είναι μια ε, ίστα της ε, ώρας ε, διακυβέρνηση. Δεν θα κάνετε αυτό το οποίο έκαναν οι Αμερικανοί ώστε να μπορέσει να αυξηθεί το ίδιο κεφάλαιο των τραπεζών, να σταματήσουν οι κερδοσκοπικές δράσεις και το συστημικό κίνδυνο να τον μειώσετε. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως είναι μια νομιμοποίηση δημοκρατική με ένα σώμα δύο κλιμάκων κοινοβουλευτικού ελέγχου ώστε να μην είναι δυνατόν να ε, να τροχοπεθηθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε κύριο Σότμαρ Κάρας. Κάρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πρώτον, η κρίση μα δείχνει με σαφήνεια τα όρια των συνθήκων και τις ε, δυνατότητές τους. Τις δικές μας ε, αδυναμίες με την διπλή ηθική θα έλεγα όσον αφορά και την απουσία κάθε σοβαρότητας από πλευρά μας. Δεύτερον, μας δείχνει σαφώς και με ανάγλυφο τρόπο ότι όποιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ο ίδιος βλάπτει τον εαυτό του αλλά βλάπτει και την ευρωπαϊκή κοινότητα. Και αυτό ισχύει για τα κράτη-μέλη πρώτον, αλλά επίσης και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτον, όποιος θέλει να ρυθμίσει στόχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν υπάρξει συμφωνία για κυρώσει, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εξαρτάται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαρτάται από την έγκριση των κρατών μελών για να κάνει τη δουλειά της. Χρειαζόμαστε αυτοματοποίηση των μηχανισμών κυρώσεων και όσον αφορά το Συμβούλιο, σταματήστε την τροχοπέδηση τη Ευρωστάτ. Πρέπει να μπορεί να ελέγχει η Ευρωστάτ τα κράτη-μέλη όποτε επιθυμεί και να μπορεί να συζητεί και να εξετάζει όποιον επιθυμεί και χρειάζεται. Πληροφορίε, ναι. Όχι όμω κάποιε ε, εκπροημίου συμφωνίε. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό είχατε κύριε. One minute. minutes. Δύο λεπτά. Λέτε. συγγνώμη, ένα λεπτό είχα εδώ μπροστά μου. Ζητώ συγγνώμη. Συνεχίστε λοιπόν παρακαλώ. Πέμπτον, λέει ο κύριος Σακάρας, θίξατε το θέμα των hedge funds, των κερδοσκοπικών ταμείων δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Πρέπει όμως ταχύτατα το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο ώστε πριν από τις διακοπές σε πρώτη ανάγνωση να αποφασίσουμε τα σχετικά. Τέλος συναλλαγών. Δεν το απαιτήσαμε όμως να το μπορέσει να υλοποιηθεί. Να δράσει η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή για το τέλος και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το τέλος επί των συναλλαγών να μπορέσει το Συμβούλιο να εξετάσει την συμβατότητα όλων των εθνικών νόμων με, το Ευρωπα... με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Χρειαζόμαστε μία μελέτη επιπτώσεων όλων των μέτρων στην πραγματική οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, λιγότερο διακυβερνητικό επίπεδο. Πρόεδρος, των διακόπτη, σας ευχαριστούμε κύριε. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Και τώρα στη συνέχεια ο κύριος Μπούλμαν παρακαλώ. Äh, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Γκαρίδο, που εκπροσωπείτε το Συμβούλιο, έχω μια πολύ συγκεκριμένη, εξειδικευμένη ερώτηση σε εσά για να μπορέσουμε από αυτή την ανικανότητα και την ανυμπόρια να μπορέσουμε να δράσουμε σε σχέση με αυτή την κρίση, να μάθουμε σε τι οφείλεται αυτή η κρίση για να την αντιμετωπίσουμε. Είμαι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος συνάδελφος Σούλτς έκανε λόγο για τα κερδοσκοπικά αυτά προϊόντα τις ασφαλίσεις και τις ασφάλειες των ε, ομολόγων και των, χρηματοπισ... των ε, μετοχών αυτών. Τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία. Γιατί κύριε Γκαρίδο και εσείς ε, συχνά είχατε συναντήσεις το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το Συμβούλιο Κοφίν. Γιατί δεν ήταν δυνατόν σε μια συντονισμένη δράση των κρατών μελών αυτά τα προϊόντα να απαγορευτούν. Εγώ την ίδια τη δική μου εθνική πρωτεύουσα ρώτησα πολύ συχνά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και χρειαστήκατε μήνες ολόκληρους ε, για να μπορέσετε να δράσετε επιτέλους. Ερωτώ, γιατί έπρεπε να πέσει πρώτα το παιδί μέσα στο πηγάδι και να κινδυνεύει να πνιγεί για να ληφθούν τα πρώτα αναγκαία μέτρα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την οικονομία μας. Και πιστεύω ότι αυτό συσχετίζεται κάπως με το ότι όταν λέτε ότι υπάρχουν αυτοί οι τρομεροί βραδύτατοι ρυθμοί, αυτή η νοσηρή βραδύτητα στο Συμβούλιο. Σας προτείνω μια συμμαχία. Εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσει. Υποβάλαμε και προτείναμε στη ρύθμιση των διοικητικών ε, επιτροπών ε, και ε, σωμάτων, στη συζήτηση με τα hedge funds και τι ρυθμίσει. Είπαμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλυφθούν τέτοια, τέτοια μέτρα και πρωτοβουλίε. Και κύριε Λάγεν, αν το κάνατε αυτό, αυτό το οποίο πάντα λέτε για τα παράγωγα, αν το αποφασίζατε, και τώρα εμείς σας το προτείνουμε και το ζητούμε κατεπηγόντως. Και λέμε, ερωτούμε και ζητούμε το Συμβούλιο επιτέλους ε, να κινητοποιηθεί, να δράσει, ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κινητοποιηθούμε. Τότε δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε αυτή την νοσηρή, απαράδεκτη βραδίτητα του Συμβουλίου. Θα έχουμε τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα που χρειάζονται για να δράσουμε. Παρακαλώ να κινητοποιηθεί το Συμβούλιο στο νομοσχέδιο θετικό επίπεδο αυτό είναι το αποφασιστικό σημείο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείτε ο χρόνος ε, αγόρευσης που έχετε και τώρα η κυρία Ντεσάρνε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι ίσω η σοβερότερη κρίση που γνώρισε η Ευρώπη. Γι' αυτό είναι επίγον θέμα. Πρέπει να λάβουμε καλέ ε, ε, αποφάσει χωρί να περιμένουμε το μήνα Οκτώβριο. Το σχέδιο διάσωση ήταν μια καλή απόφαση, βεβαίω καθυστερημένη, καλύτερα αργά παρά ποτέ, καλό αργά παρά ποτέ, αλλά θα πρέπει μακροπρόθεσμα να έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, ένα ευρωπαϊκό ομολογία, μια ευρωπαϊκή ομολογιακή αγορά και μια ευρωπαϊκή υπηρεσία αξιολόγησης βαθμολόγησης. Το ευρωπαϊκό νόμισμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σύγκληση οικονομική, φορολογική, δημοσιονομική και πολιτική διότι τότε αφήνουμε το χώρο στις αγορές και στους κερδοσκόπους. Μιλάμε πολύ για διακυβέρνηση οικονομική, αλλά θα πρέπει να συγκεντρωθούμε πάνω στο θέμα της ίδιας της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλειψε τον τελευταίο καιρό και θα πρέπει να έχουμε δύο στόχους. Ναι, βεβαίως πρέπει να μειώσουμε το χρέος, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ρεαλιστικό και με τρόπο αξιόπιστο και θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε περιθώρια ελιγμού, να έχουμε μεταρρυθμίσεις για να προετοιμάσουμε το μέλλον. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνουν τα δύο αυτά πράγματα. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα προτιμούσα να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή και είναι ζωτικό να μεταρρυθμίσουμε την φορολογία μας, να είναι περισσότερο στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, να την εναρμονίσουμε. Δεν θα έχουμε νομισματική ένωση χωρί δημοσιονομική, οικονομική και πολιτική κυρία Πασκάλ Καντιέ. Ο κύριος, με συγχωρείτε. Mm. Κύριε Ρέν. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να μειώσει κανείς τα ελλείμματα. Η μείωση των δαπανών και η αύξηση των εσόδων. Όλοι μπορούν να περικόψουν τις δαπάνες ταυτόχρονα ή ξεχωριστά. Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκό συντονισμός γι' αυτό. Να αυξηθούν τα έσοδα, τα φορολογικά, φορολογία πάνω ε, στο κεφάλαιο, στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συντονισμός ευρωπαϊκός και στην ανακοίνωσή σας την περασμένη εβδομάδα δεν αναφέρεται τίποτα για το θέμα αυτό. Η ερώτησή μου η οποία την συμμερίζονται πάρα πολλοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανεξαρτήτως των ομάδων είναι στις επόμενες εβδομάδες θα έχετε ένα σχέδιο ε, φορολογικής δημοσιονομικού συντονισμού για να έχουν τα κράτη-μέλη να ξαναβρούν περιθώρια λιγμού για να αυξήσουν ορισμένους φόρους, πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν ξεχωριστά. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα. Δεν είδα τίποτα. Ο κύριος Φερχοφστάντη είπε έχετε δικαίωμα πρωτοβουλία. Σήμερα έχετε καθήκον πρωτοβουλία ως προς τον τομέα. Σα ε, Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαντάλε Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, φοβούμε ότι δεν θα λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα. Καμιά χώρα παγκόσμια δεν το κατάφερε ένα τέτοιο τεράστιο έλλειμμα μέσα σε τρία χρόνια να το μειώσει και η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις κατά των μέτρων λιτότητας. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, να περάσει σε μια σπυροειδή εξέλιξη προς τα κάτω αυτή η χώρα με μειούμενες ε, δαπάνες. Χρειάζονται όμως περισσότερες ε, δημόσιες δαπάνες ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι τόκοι και οι πιστώσεις. Θα πρέπει να κρούσουμε κόδωνα κινδύνου. Κάποτε πρέπει να αναφερθεί. Υπάρχει κίνδυνος εδώ εξόφλησης των χρεών. Και τι γίνεται δεν γινόταν λέει διαφορετικά. Κάποιες τέτοιες δηλώσεις ακούμε. Και τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να τηρήσουν τα υπεσχημένα οι χώρες, τα κράτη-μέλη χρειάζονται ε, πραγματικά έντιμα στοιχεία τα οποία θα διαθέτουν και θα διαβιβάζουν. Πρέπει να εξηγιανθεί η κατάσταση, να, να αποπληρωθούν τα χρέη. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την κατάσταση όσο έχει. Ο κύριος Νικόλαος Χουντής παρακαλώ. Πρόεδρε αύριο στην ελλάδα θα γίνει η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση της τελευταίας δεκαετίας οι έλληνες εργαζόμενοι αντιστέκονται στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση εργαζόμενοι που ούτε δουλεύουν λιγότερο ούτε αμείβονται καλύτερα από τους άλλους συναδέλφους παρακαλώ κοιτάξτε τα στοιχεία. κύριε ρεν αποτελεί μέγιστη υποκρισία όταν αυτό το μηχανισμό της τριμερούς χρηματοδότησης τον ονομάζεται μηχανισμό σωτηρίας και αλληλεγγύης. πρόκειται για μηχανισμό ευρωπαϊκής τιμωρίας με το διεθνές νομισματικό ταμείο στο ρόλο του κακού. επί έξι μήνες σας προτείναμε να αξιοποιήσετε το άρθρο 122 ε, της συνθήκης της λισαβόνας. επί έξι μήνες καλούσαμε την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να αλλάξει πολιτική. επί έξι μήνες σας καλούσαμε να ελέξετε τους απαράδεκτους αμερικάνικους οίκους αξιολόγησης. δεν το κάνατε. αφήσατε να κάνουν πάρτι οι κερδοσκόποι φέρατε το διεθνές νομισματικό ταμείο στην ευρωζώνη τώρα ζητάτε σκληρά ε, προγράμματα λιτότητας. αυτό το μηχανισμό πρέπει να το συζητήσει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 της συνθήκης της λισαβόνας και πρέπει να συζητηθεί πραγματικά μια πολιτική αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε. <clears throat> παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε με την πομπόδη παρουσίαση από πλευρά τη Ισπανική Προεδρία θυμόμαστε το ότι ακούσαμε τώρα, όμω ε, μετά από την Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ 11% ε, του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία αμέσω ψάχνει να βρει κάποιον ε, να θεωρηθεί υπεύθυνο. Το γεγονό όμω είναι ότι αυτή η γραφειοκρατία είναι υπεύθυνη για αυτήν την κρίση, διότι έβαλε κράτη στην ζώνη του ευρώ γνωρίζοντας ότι οι οικονομίες τους ε, δεν ήταν υγιείς. Και πόσες χιλιάδες απασχολούνται στην ε, Ευρωστάτα. Απλά και μόνο συλλέγουν στοιχεία, τι κάνουν. Και κάποιοι υποφελούνται από την ε, κατάσταση. Όμως δεν δημιούργησαν αυτή την κρίση. Τώρα ζητούνται μειώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ρεαλιστικό αυτό σε σχέση με το δημόσιο κόστος στην Ελλάδα να μπορέσει να αναμένεται αυτή η εξέλιξη όταν υπάρχουν τόσοι που εργάζονται στο δημόσιο. Και τώρα ένα πακέτο μέτρων διάσωσης ε, έχει υιοθετηθεί. Όμως ε, θα πρέπει να συνεισφέρουν ε, χώρες που δεν έχουν τα χρήματα να συνεισφέρουν. Το ίδιο γίνεται και σε σχέση και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόεδρος διακόπτη, συνάδελφε, πρέπει να σας διακόψω. Μόλτσερ, δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, υπερβολικά γρήγορη κεντρική διακυβέρνηση και ίσως ε, σε σχέση με τα μέτρα τα οποία λήφθησαν ήταν συνυπεύθυνα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σήμερα. Ευρωπαϊκό νόμισμα το οποίο δεν μπόρεσε μακροπρόθεσμα να μπορέσει να ε, ευδοκιμήσει διότι είχαμε ένα ε, σύμφωνο το οποίο δεν ήταν λειτουργικό. Και τώρα λέμε ότι πρέπει να υπάρξει κοινή κεντρική οικονομική διακυβέρνηση. Κάτι σαν μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Είναι σωστό όταν έχουμε ε, χώρες που είναι αδύναμες και θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη πρέπει να υποστούν αυστηρότατους ελέγχους ε, όσον αφορά τις πολιτικές τους. Όμως μια κεντρική διαμόρφωση των πραγμάτων με τις Βρυξέλλες ως το επίκεντρο θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτη ανάμειξη στην, στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Αυτό θα σήμαινε πραγματικά να θελήσουμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια με άλλη ασθένεια. Και έτσι εδώ δεν είναι δυνατόν σε σχέση με τις ε, Επιθυμίε που έχουμε σε κεντρικό επίπεδο να τι διαμορφώσουμε. Σε σχέση, για παράδειγμα, με τη συνθήκη της Λισαβόνας, αν θέλουμε να συναγάγουμε μαθήματα από τη σημερινή κρίση, ίσως μια τελείω άλλη διαφορετική δομή και διάρθρωση θα χρειαζόμαστε για την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική. Κάτι σαν ένα σκληρό κεντρικό νομισματικό πυρήνα. Ε, μια ε, κεντρική, θα έλεγα, ενωμένη Ευρώπη που θα έπρεπε να δράσει ώστε να μπορέσει να εξηγιαθεί προγράμματα λιτότητας θα πρέπει να είναι στο μέλλον ο κανόνας και το γνωρίζουμε αυτό. Είναι σαφές όταν τα κράτη πρέπει να ε, εξοικονομήσουν, οι πολίτες να εξοικονομούν ε, με τις πολιτικές που τους επιβάλλονται, τότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική λιτότητας. Πρέπει εδώ λοιπόν να είμαστε σοβαροί στα δημοσιονομικά μας και πρέπει να εξετάσουμε και εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο σε περίοδο δημοσιονομικής πειθαρχίας και περικοπών να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα γραμματείας ε, και αρρωγής που δίνεται στους ευρωβουλευτές για τους βοηθούς. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Την ημέρα εκείνη όπου είχαμε την επέτειο των 60 ετών από την διακήρυξη Σούμαν, το Συμβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενταφίασε την μέθοδο του Μονέ για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν τα νομικά πλαίσια σε σχέση με την κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων. Τα δέχτηκε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με τις επικρίσεις του συναδέλφου Φεχόστατ δεν είναι ε, κρίση του συστήματος και του ευρώ, είναι κρίση των κυβερνήσεων. Και όταν βλέπουμε ότι έχουμε εδώ την, τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας, τι έκανε η Ισπανική Προεδρία πρέπει να ρωτήσω. Ούτε ιδέες συνεισέφερε, ούτε πρωτοβουλίες ανέλαβε. Και εδώ συζητούμε το σοβαρότατο πρόβλημα της Ευρώπης ε, σήμερα. Και ε, σε σχέση με τη Σύνοδο της Μαδρίτης, τι είναι εκείνο το οποίο ζητείτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχτηκε όλα όσα προτάθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άφησε το Συμβούλιο να την χειραγωγεί και μετά από πάρα πολύ σοβαρές προσπάθειες μόνο μία ανακοίνωση δημιουργήθηκε. Μόνο μία ανακοίνωση ήταν το προϊόν. Έχει δίκιο ο συνάδελφος Μπούλμαν. Πού είναι οι συγκεκριμένε εξειδικευμένες προτάσεις εδώ χρειαζόμαστε προτάσεις για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Δεν επαρκούν αυτά τα οποία έγιναν. Θέλουμε να έχει θάρρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την μέθοδο την κοινοτική, την μέθοδο του Ζαν Μονέ, υπέρ των θεσμικών οργάνων, υπέρ κοινοτικών προτάσεων που θα υποβληθούν. Και όλοι ξέρουμε ότι η συνεργασία των κρατών μελών σε οικονομικά και νομισματικά θέματα πρέπει να διασφαλίζεται. Αυτό είναι το αίτιο, η αιτία αυτή τη κρίση. Ότι δεν συμμετείχαν τα κράτη-μέλη και δεν συνεργάστηκαν. Και έκαναν κιόλα και παρεκκλήσει, ε, οδηγήθηκαν σε παρεκκλήσει. Και μπορώ να πω σε ένα σημείο ότι ο συνάδελφο Σούλτ δεν μίλησε εδώ <clears throat> σαν ο ηγετικός ε, ρόλος ε, της ε, ομάδας του να ήταν ο μόνος δεδομένος. Όμως ένα σημείο έχει δίκιο και εμείς εκφράσαμε το παράπονο ότι οι Έλληνες συνάδελφοι από τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το πακέτο στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν το υποστήριξαν. Αυτό είναι κάτι το ανεύθυνο πιστεύω εγώ. Όμως υπάρχει το δικαίωμα να επισημανθεί ότι όλες οι κρίσεις και όλα, όλοι όσοι έχουν τροχοπεδίσει τα πράγματα σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία την Ουγγαρία, την Ισπανία με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει υπευθυνότητα εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Λόπες Αγγιλιάρ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε τη θητεία μας ε, και σε κάθε ολομέλεια ε, συζητάμε την κρίση. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια κρίση που μείωσε τρομερά την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δεν θέτουμε σωστά την εξίσωση δεν πρόκειται να τη λύσουμε. Η κρίση δεν αφορά το ευρώ και την Ελλάδα μόνο, αλλά έδειξε ανισορροπίε που είναι αβάσταχτες και θα πρέπει να τι ε, αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, διαφορά ανάμεσα στην οικονομική και στην, πραγματική, ε, στην χρηματοπιστωτική και στην πραγματική οικονομία. Δεύτερον, ύπαρξη νομισματική Ένωση, αλλά έλλειψη οικονομική Ένωση, φορολογική Ένωση. Ε, ε, ε, που να μπορεί να συνοδεύει τι απαιτήσει τη Νομισματικής Ένωση. Τρίτον, η ένταση τη κρίση, οι τρομερέ προκλήσει και η αβάσταχτη βραδύτητα απόκριση που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και του θεσμού. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του άνεργου, στρατιέ των άνεργων που έχουν τα βλέμμα, το βλέμμα του στραμμένο επάνω μα. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Κοιτάξτε, είδα από τη μια ε, από αποφάσεις όσον αφορά ε, το, ε, το περασμένο Σαββατοκύριακο της, ε, της Συνόδου Κορυφής. Και έχουμε και τη στρατηγική 2020. Αλλά κοιτάξτε, αυτές οι αποφάσεις, μην το ξεχνάμε, ότι συνοδεύονται από τρομερές απαιτήσει από τις χώρες που δεν μπορούν να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Άρα λοιπόν και αυτό μπορεί να σημαίνει αναχέτηση της ανάπτυξης. Κοιτάξτε, χτε μιλούσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μιλούσαμε για το πρόγραμμα δράση του προγράμματο Στοκχόλμη. Επ' ευκαιρία λοιπόν αυτή τη συζήτηση ε, ε, θυμηθήκαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη δεν είναι μόνο η οικονομική ένωση, δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο συγγνώμη, νομισματική ένωση, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά αλλά και του πολίτε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών εκφράζουν τη δυσαρέσκειά του απέναντι στην Ευρώπη που του προσφέρουμε. Αυτή την Ευρώπη που εκτοξεύει απειλέ ε, ε, και τιμωρίε προ τι χώρε που δεν εκπληρώνουν τι υποσχέσει του, αλλά δεν αντιμετωπίζει τι δικέ δεσμεύσει για απασχόληση, για κοινωνική συνοχή, για τα καταπολέμηση τη φτώχεια. Χωρί αυτή την, την Ευρώπη των πολιτών δεν πρόκειται να επιληθεί και η συγκεκριμένη κρίση. Κύριε για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον Επίτροπο και την Ισπανική Προεδρία για όσα έγιναν ε, πρόσφατα ακόμα και καθυστερημένα. Δεν είναι εύκολο κανείς ε, να κυβερνά όταν υπάρχει θύελα. Κάνατε σε 14 μέρες πολύ περισσότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και θα ήθελα να συνεχίσετε. Ένα μήνυμα στην Ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να πω ότι το μήνα Ιούνιο θα είστε υπεύθυνοι για την υιοθέτηση της στρατηγικής 2020. Μην υιοθετήστε κάτι ε, που να μην αξίζει η στρατηγική της Λισαβόνας δεν λειτουργήσε καλά τα περισσότερα προβλήματα προέρχονται από την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις χώρες του Νότου το είπε ο κύριος Βέρχοφστατ χρειαζόμαστε ε, χρηματοοικονομική παρακολούθηση επιτήρηση είμαι εισηγήτρια για τον συστημικό κίνδυνο ε, νομίζω ότι η λέξη συστημικός επαναλήφθηκε πολλές φορές τι τελευταίες εβδομάδες έχετε την ευθύνη αυτού του πακέτο να είστε φιλόδοξοι, έχετε την υποστήριξή μας. Μην ακούτε αυτούς στο Συμβούλιο που θέλουν να μην υπάρχει ρύθμιση. Για τον κύριο Ρεν, του οποίου χαιρετίζω το θάρρος, υποστηρίζω πλήρως το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει στα Εθνικά Κοινοβούλια να συνεργαστούν στην ε, πηγή, στα ανάντι με τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά ε, να μην υπάρχει για όλους τους λαϊκιστές εδώ μια ευκαιρία και για όσους κατακρίνουν την Ευρώπη. Έχετε την υποστήριξή μας, αλλά προσπαθήστε να συνεργαστείτε καλά με τα εθνικά κοινοβούλια και να μην δίνετε την εντύπωση ότι οι Βρυξέλλες υπαγορεύουν στα εθνικά κοινοβούλια τι πρέπει να κάνουν. Τα εθνικά κοινοβούλια που είναι θεματοφύλακες της δημοκρατίας έβαλαν την Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση ψηφίζοντας τέτοιους ελληματικούς προϋπολογισμούς εδώ και χρόνια και χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία μας έφεραν οι κυβερνήσεις μας. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι έλειπαν οι κανόνες για την αποφυγή της κρίσης. Ε, εάν υπήρξε συμφωνία με τα κριτήρια του Μάστερ με, το, Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, δεν βρισκόμασταν σε αυτό το επίπεδο κρίση το οποίο ε, αντιμετωπίζουν πολλά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ε, βρίσκομαι στην παράδοξη κατάσταση να μιλώ ε, ε, για τις ε, ε, επενδυτικές τράπεζες και για τις οικονομικές δεξιότητες των κρατών μελών. Κάθε φορά μιλάμε για τις τράπεζες, για το γεγονό ότι δεν υπακούν στους κανόνες, ότι ακολουθούν διάφορα τεχνάσματα. Μα αυτό ακριβώ κάνουν και οι κυβερνήσει. Ζητάμε ε, ε, εταιρική διακυβέρνηση υπεύθυνη. Ε, έχουμε φτιάξει διάφορα μέσα ε, αντιμετώπιση ε, επίγουσων κατα... αναγκών κτλ. Και όμω ταυτόχρονα οι κυβερνήσει δεν έχουν σταθεί στο ύψο ε, των περιστάσεων και δεν έχουν δείξει την υπευθυνότητα που θα έπρεπε. Αυτό έγινε και στη χώρα μα και το ανακαλύψαμε αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε ε, την κατάσταση των οικονομικών στη χώρα μα. Αυτό πρέπει να κάνουν και, και οι άλλε χώρε μέλη και να βρουν έναν τρόπο για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. για ένα λεπτό. Πρόεδρε, μια συντονισμένη πολιτική για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι απόλυτα αναγκαία. Όμως ε, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε τα μεγάλα θεσμικά όργανα. Τα χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα έπρεπε να διασωθούν επειδή δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους ε, τα τελευταία δύο χρόνια. Στην Ολλανδία τι έγινε. Στην Ολλανδία έπρεπε να πληρώσουμε 2,5 δις ευρώ επιπλέον όσον αφορά πληρωμές τόκων και <clears throat> το Ταμείο Συντάξεων έπρεπε να πληρώσει ένα δις ευρώ όσον αφορά την αγορά ε, ομολόγων και σε, με πολύ υψηλά επιτόκια και υπάρχει κερδοσκοπική δράση. Πρέπει να σωθούν λοιπόν αυτά τα, να σωθεί αυτό το Συνταξιοδοτικό ταμείο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα αναγκαία μέτρα, όχι σε ακραία μέτρα, αλλά να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και να αναχαιτήσουμε τις κερδοσκοπικές τάσεις ε, που είχαν τόσο αρνητικές επιπτώσεις στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν το σωστό πρότυπο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω απόλυτα σε θεωρητικό επίπεδο τις προτάσεις του κυρίου Όλι Ρεν, τον οποίον τολμώ να θεωρήσω πολιτικό κεφάλαιο για την Ευρώπη και ε, πρόσωπο στο οποίο πρέπει ιδιαιτέρως να αποδίδουμε τιμή. Εκείνο το οποίο όμω θέλω να πω και να επισημάνω ότι ο μεγάλος πυρετός είναι εξίσου επικίνδυνος με την υποθερμία και στην οικονομία και στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και στην οικονομία. από τη βραδία προσαρμογή του μάστριχ η οποία πέρασε για πολλά χρόνια και ε, όλη η οικονομία της ευρώπης δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στην αναγκαστική και βίαιη προσαρμογή που θα οδηγήσει σε μια παράταση της ύφεσης. οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω ότι η παγκόσμια οικονομική αταξία που συνεχίζεται οφείλεται κυρίως στη δημιουργία μεγάλων αζήτητων αποθεμάτων ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ε, προσπάθεια τόνωσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο της ανάπτυξης εις τρόπον ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ορθολογικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Κίφερ Χόφστας κατήγγειλε την ανεπάρκεια των ρητορικών, εθνικιστικών και μαρξιστικών ε, ως τρόπο για να ξεφύγουμε από την κρίση. Ε, για να προσπαθήσω λίγο με τη ρητορική, την ευρωπαϊκή θα έλεγα. Πριν από λίγε εβδομάδε σε αυτή την αίθουσα, πολλοί από εμά αναφερθήκαμε στο θέμα τη αλληλεγγύη υπέρ της Ελλάδας. Σε τι χρησιμεύει λοιπόν η Ευρώπη εάν δεν μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη όταν βρίσκονται, όταν αντιμετωπίζουν ε, συγκεκριμένε ανάγκε. Σε τι χρησιμεύει το ευρώ και, το, και η ευρωζώνη εάν δεν προωθούν μία, μία νοτροπία ευθύνης και σταθερότητα, τι θα συνέβαινε για πράγμα, πράγματι εάν η αλληλεγγύη ε, γίνει συνώνυμο μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παραβιάζει τι συνθήκε ε, και τελικά ε, από τη μια έχουμε τις, τα κράτη-μέλη τα οποία θυσιάζουν το, το μέλλον των ίδιων των πολιτών, αν θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Ρητορική Επίτροπε σημαίνει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τι ευθύνε τη και να αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη τα οποία παραβιάζουν παραβιάζουν τις, ε, τους ε, κανόνες, ε, που φροντίζει για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, που, μειώνει, που προσπαθεί να μειώσει τα σφάλματα στην οικοδόμηση του ευρώ. Όταν δηλαδή δεν έχουμε και αντιμετώπιση των φόρων και των συντάξεων, για παράδειγμα. Ναι, είναι αλήθεια, βρισκόμαστε σε μια κρίση. Αλλά η κρίση αυτή δεν προήλθε από υπερβολική Ευρώπη. Αντίθετα, προήλθε από ανεπάρκεια της Ευρώπης. από πολύ λίγη Ευρώπη, αν θέλετε. Μία Ευρώπη που θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να λάβουν τις ευθύνε τους, να, να φροντίσουν τη σταθερότητα, το μέλλον των επόμενων γενεών. Και όλα αυτά δεν είναι ρητορική. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα γίνουν πραγματικότητα, θα εφαρμοστούν στην πράξη. Δηλαδή θα αποτελέσουν μέρος μιας πολιτικής στρατηγικής που θα, προλα... που θα προλαβαίνει τα γεγονότα και που δεν θα προσπαθεί να μειώσει τις συνέπειες. Ο κύριος Σασόλη για δύο λεπτά. Europa dei popoli e non una μια Ευρώπη λαών και όχι Ευρώπη των κρατών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η κρίση που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι ε, κρίση μια ευρωπαϊκή πολιτική που κατέστη ανίκανη να ε, φροντίσει για τη διακυβέρνηση των αγορών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικοί θεσμοί, να βγούμε από τη διακυβερνητική λογική και να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτά δεν είναι ρητορική. Γιατί πριν από λίγα λεπτά ε, στο Βερολίνο η Γερμανίδα καγκελάριο, η κυρία Μέρκελ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και είπε ότι το ευρώ ε, βρίσκεται σε κίνδυνο. Μάλιστα, το να, το το να κινδυνολογούμε όμω χωρί να φροντίζουμε έτσι ώστε να ληφθούν ε, πιστικά μέτρα απέναντι στου επενδυτέ, απέναντι στην αγορά, ε, τελικά αποδυναμώνουμε ακόμα περισσότερο το ενιαίο μα νόμισμα. Ε, ε, και με αυτόν τον τρόπο καθιστούμε πιο αδύναμη ολόκληρη την Ευρώπη. Για να φανταστούμε ε, την, την απάντηση των αγορών όταν δηλαδή πριν από λίγα λεπτά βλέπουμε τι γίνεται με το ευρώ και πώς πέφτει για άλλη μια φορά. θα, θα βρεθούμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι πιο φτωχοί και, και ακόμα περισσότερο ανασφαλείς. Μόνο μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση θα μας βοηθήσει να υπερασπιστούμε το ενιαίο μας νόμισμα, να προωθήσουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ε, ενσωμάτωση και ένταξη. Ας ξεχάσουμε την προσέγγιση μέσα από εθνικές πολιτικές. Ας φροντίσουμε να έχουμε ισχυρά μέσα λήψη αποφάσεων μέσα από τρία επίπεδα παρέμβασης. Πολιτική για την ανάπτυξη, ε, σωστά χρηματοπιστωτικά μέσα, διαχείριση των έκτακτων αναγκών ε, ε, όσον αφορά αυτό το σχέδιο των 750 δις είναι σημαντικό αλλά από ό,τι καταλάβαμε δεν αρκεί. Σήμερα χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική πρωτοβουλία γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ε, θα καθοδηγήσουμε τις αγορές και θα πετύχουμε υψηλή κινητοποίηση των πόρων σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, σε νομισματικό επίπεδο γιατί τελικά δεν, δεν έχουμε μπορέσει μέχρι στιγμής να εγγυηθούμε την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Μη φοβόμαστε την ανάπτυξη κυρίως σε σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος, ενέργεια, περιβάλλον, γνώση, ε, ανθρώπινο κεφάλαιο. Το κοινοβούλιο μας, ε, κύριε Πρόεδρε, έχει ε, πολύ μεγάλες ευθύνε. Θα πρέπει να ενισχύσει με τη δική του την ανεξαρτησία και την αυτονομία, την ικανότητα των κρατών έτσι ώστε να μπορέσουν να φύγουν από τη διακυβερνητική λογική και να ακολουθήσουν το δρόμο του ευρωπαϊκού πνεύματος. και κύριοι, οι αγορές ε, οδηγούν τις ε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυτές αντιδρούν, αντιδρούν εκ των υστέρων, δεν δρούν ε, εκ προημίου. Είναι σκάνδαλο, σκανδαλώδες ότι οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρούν όταν δείχνουν τις αδυναμίες τους οι αγορές. Έπρεπε όμως ε, να έχουν αναγνωριστεί έγκαιρα αυτές οι αδυναμίες. Ε, όταν εισήχθη το ευρώ γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε το χρήμα εκείνο το οποίο απαιτείται από τα κράτη-μέλη και λάβαμε μέτρα για να υπάρξει υποκατάστατο. Όμως δεν τηρήσαμε αυτά τα μέτρα και μάλιστα μεγάλα κράτη-μέλη σαν του κανόνε. Χρειαζόμαστε αυστηρέ ρυθμίσει και μηχανισμού ε, να ονομάζουμε, να κατονομάζουμε και να επικρίνουμε αυτού ε, που, να κατακρίνουμε αυτού που δεν τηρούν τα υπεσχημένα. Δεύτερον, είναι σαφέ ότι έχουμε εσωτερικέ εντάσει στην Ευρωζώνη που οδηγούν σε μια πραγματική κρίση βιωσιμότητα επειδή έχουμε διαφορετική ανάπτυξη και διαφορετική ανταγωνιστικότητα. Εδώ πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Πρέπει οι προπολογισμοί των επιμέρου κρατών ε, να μπορέσουν να εξεταστούν και να δούμε αν υπάρχει κίνδυνο για την Ευρωζώνη από αυτή την κατάσταση. Φυσικά ξέρουμε ότι τα ε, νομισματικά και ε, δημοσιονομικά δικαιώματα είναι κυρίαρχα δικαιώματα των κοινοβουλίων, των κρατών μελών. Όμω εδώ χρειάζεται κατεπηγόντω περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Αυτό είναι πραγματικά η τελευταία μα ευκαιρία. Αν εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν δράσουν από κοινού με το Ευρωκοινοβούλιο, τότε θα υπάρξει τεράστια ζημιά που θα υποστούμε όλοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν ότι δεν υπάρχει επαρκής Ευρώπη για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης εκείνο το οποίο μας ε, απασχόλησε ήταν ε, η ρύθμιση θεσμικών θεμάτων. Αγνοήσαμε όμως ε, την συνεργασία και τον συντονισμό στην καταπολέμηση της κρίσης. Και εδώ καλείται αλληλεγγύη να υπάρξει στην καταπολέμηση της κρίσης. Για παράδειγμα, όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία, υπάρχουν εκεί πάμπολοι οι οποίοι υφίστανται τις επιπτώσεις αναμένουν και προσδοκούν ότι κάτι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βλέπουν να γίνονται πολλά πράγματα. Είναι αδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια ώστε να ληφθούν δημοσιονομικά μέτρα. Δεν υπάρχει λοιπόν, α το πω έτσι, ύπαρξη οικονομικών μέτρων που να ακολουθούν στόχου για την αντιμετώπιση τη κρίση. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνο να είμαστε ακόμα πιο αποδυναμωμένοι και να πληγούν οι πιο αδύναμοι. Ευχαριστώ.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έφτασε η στιγμή της αλήθειας, της οξυδέρκειας, της υπευθυνότητα αυτή την κρίση που δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή αλλά παγκόσμια. Η ε, διακυβέρνηση του πλανήτη διαμορφώνεται. Ποια θα είναι η επιρροή των Ευρωπαίων, πώς θα την επηρεάσουμε αν δεν είμαστε ικανοί να έχουμε τη δική μας ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Μετά από 50 χρόνια οικοδόμησης, ποιος δεν είδε ότι είχαμε τον κίνδυνο από διάλυση διάλυσης, διάλυσης μετά από αυτό. Έχουμε ηθαγένεια χωρίς τους πολίτες. Έχουμε εκλογές χωρίς τους ψηφοφόρους. Ένα κράτος δικαίου το οποίο δεν, το σεβόμεθα. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου επανενώσαμε την ήπειρό μας αλλά δεν είδαμε τις αδυναμίες μας. Και τώρα η κρίση μας πλήττει όλους και η ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι βάλωτο με κράτη τα οποία είναι ε, διεφθαρμένα, που είναι κακοδικούμενα και ξέρουμε όλοι ότι η δύναμη ε, μιας αλυσίδας είναι η δύναμη του πιο αδύνατου κρίκου. Πρέπει Τώρα και αυτή θα είναι η δύναμή μας να σώσουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Δεν είναι οι κανόνες οι ευρωπαϊκοί που είναι οι κακοί, είναι η εφαρμογή τους από τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν παρακολούθησε, δεν επετήρησε αρκετά τα κράτη που είχαν ελλείψεις. Μας χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, Ευρώπη αλήθειας, οξυδέρκειας, ε, διαφάνειας. Πρέπει να τηρήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που πρέπει να ανανεωθεί και να ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό περνάει από την ανάπτυξη και την απασχόληση και από την επένδυση. Αν ο δημόσιο τομέα δεν επενδύει, δεν θα επενδύσει και ο ιδιωτικό τομέα. Προτείνω λοιπόν στα 10 χρόνια της εφαρμογής της στρατηγικής 2020 100 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις ώστε το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει το πιο ανταγωνιστικό με υποδομές, με δίκτυα, ε, με τρένα υψηλής ταχύτητας, με το είδωρ, με την υγεία, την ε, παιδεία, αναμορφώνοντας ε, τους προϋπολογισμούς μας με όλους τους παράγοντες, τους δημόσιους και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κυρία Φερέρα. Eh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όταν η Οικονομική και Νομισματική Ένωση συμπλήρωσε τη δεκαετία της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε το ευρώ στο πιο επιτυχημένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Σήμερα όμως ε, ε, έχουμε κάποιες δυσκολίες γιατί βλέπουμε τους περιορισμούς του και η κρίση έδειξε ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι ένα σχέδιο που έμεινε ατελέ. Έχουμε μια κατεπίγουσα κατάσταση και δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Οι συνθήκες πίεσης και τα άμεσα συμφέροντα των βασικών χωρών μελών, ο επώδυνος χαρακτήρας των αποφάσεων, οι κολυσιεργίες στην εφαρμογή τους, κατέστησαν πιο έθραυστη την εικόνα του ευρώ και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες και στον κόσμο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι διαδικασίε ολοκλήρωση, όχι απλή ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών. Έμεινε ατελή αυτή η διαδικασία και μάλιστα διατρέχει και σημαντικό κίνδυνο εξαφάνιση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τρία θέματα πρώτα απ' όλα. Καταρχήν, είναι σημαντικό να εμπεδώσουμε τους μηχανισμούς, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό τομείο, να δημιουργήσουμε ευρωομόλογα, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ευρωπαϊκής Ρύθμιση και εποπτείας και επίση να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων. Δεύτερη διάσταση. Δεν νοείται ισχυρό νόμισμα με αδύναμη οικονομία. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και τη δημογραφική σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσπάθεια καταπολέμησης της ενεργείας. Η στρατηγική του 2020 είναι ένα σύνολο αγαθών προθέσεων και ωραίων ιδεών, αλλά χωρίς αμέσα για την υλοποίησή τους. Τρίτη διάσταση η φορολογική και δημοσιονομική εξυγίαση που είναι σημαντική αλλά δεν μπορεί να συνεπάρχει με όλο και μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των χωρών που συνθέτουν την Ένωση. Η πολιτική σύγκληση θα πρέπει να επανεξεταστεί επιγόντως. Ευχαριστώ. Ε, για λεπτό. Ήδη για τρίτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το δεκαετές σχέδιο που έχει τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη του 2020». Υπήρξε δυσφορία σε πολλούς ευρωβουλευτές, όχι μόνο επειδή κάναμε συνειρμούς με διάφορους, διάφορα πολιτικά συστήματα, αλλά εξαιτία και της παταγώδους αποτυχίας ε, της προηγούμενης συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά την τελευταία συζήτηση προτεραιότητας, επέστε την προσοχή σας στο γεγονός ότι Ορισμένα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση τη Ένωση. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έλαβαν συγκεκριμένε αποφάσει προκειμένου να σταθεροποιήσουν τη ζώνη ευρώ και τι οικονομίε των ευρωπαϊκών χωρών. Και μάλιστα η, υποσχόμενη έγχυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ θα βοηθήσει κάποιε χώρε τη Δυτική Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα. Αυτό όμω θα πρέπει να γίνει εις βάρος των χρηματοοικονομικών συστημάτων στήριξης των νέων χωρομελών, μεταξύ άλλων της Πολωνίας, που δεν ασχολήθηκαν αδιάφορα και ανέμελα με τους οικονομικούς δείκτες. Αν διατηρηθεί η στρατηγική του 2020, θα πρέπει να αποκατασταθεί μια ισορροπία σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. για λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η χειρότερη κρίση που μπορούμε να βιώσουμε δεν είναι η σημερινή. Αλλά η κρίση που θα υποστούμε αν δεν καταφέρουμε να αντλήσουμε τα σωστά πολιτικά διδάγματα σε σχέση με την παρούσα κρίση. Γιατί φαίνεται ζήσαμε πέραν των δυνατοτήτων μας σε πολλές χώρες. Απομακρυνθήκαμε από την πραγματική οικονομία και εγκολποθήκαμε την εικονική οικονομία, την φαντασία, τη φανταστική οικονομία. Και μάλιστα αυτό φάνηκε και στους κρατικούς λογαριασμούς αλλά και στους λογαριασμούς των οικοκυριών. Δεν καταλάβαμε ότι ένας ζωντανό οργανισμός ε, θα πρέπει να αναπτύσσεται, όχι να παχαίνει κατά ανάγκη. Χρειάζεται λοιπόν η ανάπτυξη, μια προσπάθεια αλλά και μια αναλογία, ενώ το υπάχυνση δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ της προσπάθειας που καταβάλουμε και της ευημερίας που απολαμβάνουμε η κρίση αυτή είναι δυναμική και το στιγμιότυπο της κρίσης πριν από μερικούς μήνες είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα της κρίσης σήμερα. Και μάλιστα η κρίση σε μερικούς μήνες είναι πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Η κρίση ήταν οικονομική και χρηματοπιστωτική και θα έχει όλο και μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση, διάσταση κοινωνικής αντιπαράθεσης και πριν περάσουμε στη φάση της κοινωνικής αντιπαράθεσης θα πρέπει εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική να συνειδητοποιήσουμε ότι η βασική κρίση είναι κρίση συνείδη, ε, εμπιστοσύνης και όχι μόνο κρίση του ευρώ. Θα πρέπει να αναλύσουμε όλα τα πολιτικά μας συστήματα, γιατί υπάρχει σημαντική κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιες αλλαγές θα πρέπει να επιφέρουμε, τι αλλαγή νοοτροπίας θα πρέπει να γίνει, τι αλλαγή πολιτικής, θεσμικής, προσωπικής νοοτροπίας. Και από αυτή την άποψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντί να σκέφτεται άλλα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να διαρωτηθεί ποια μπορεί να είναι η συμβολή μας προκειμένου να αλλάξει η θεσμική και πολιτική νοοτροπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σήμερα άκουσα πολλούς λόγους για την κρίση. Τη γραφειοκρατία, τους οργανισμούς αξιολόγησης, τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν όμως δύο ζητήματα στα οποία θα πρέπει να επιφέρουμε αλλαγές. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μια συνοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να χάνουμε τις δυνάμεις μας και να λανόμαστε σε μια τόσο ευρυθή συζήτηση για τη διάσταση της κρίσης και θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, την αλήθεια για αυτό που μας συμβαίνει. Ευχαριστώ. πρώτα απ' όλα συμπληρωματικά δέκα δευτερόλεπτα θα ήθελα να σας παρακαλέσω επί του διαδικαστικού και για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας είπε πριν ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος λάγκεν δεν είναι τώρα στην αίθουσα χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι έλληνες συνάδελφοι καταψήφισαν το τριετές πρόγραμμα σταθεροποίησης στο ελληνικό κοινοβούλιο και ήθελα να σημειώσω ότι ε, θα ήταν καλό ο κύριος λάγκεν να επαναλάβει αυτές τις συστάσεις στο πλαίσιο της επόμενης συνόδου του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος γιατί στο ελκ ανήκουν αυτοί οι συνάδελφοι που όλο τυχαίω είχαν και την ευθύνη τη διακυβέρνηση τη χώρα μέχρι πριν από λίγου μήνε. στο γενικότερο θέμα τώρα κύριε πρόεδρε είναι γεγονό ότι η σημερινή κρίση έφερε στο προσκήνιο μόνιμε παθογένειε και αδυναμίε και σε ό,τι αφορά στον οικονομικό συντονισμό τη ευρωζώνη αλλά και στο παγκόσμιο σύστημα οικονομική διακυβέρνηση με αποτέλεσμα να σωρεύονται τεράστιε ανεξέλεγκτε εξουσίε στο παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχουμε λοιπόν σήμερα πρώτα και πάνω απ' όλα ένα ζήτημα δημοκρατίας να αντιμετωπίσουμε και η ευρώπη αν θέλει να σεβαστεί τις αξίες και την ιστορία της πρέπει πρώτα να πρωταγωνιστήσει στην υπόθεση αυτή. η απόφαση για τη συγκρότηση ενός μηχανισμού στήριξης της σταθερότητας της ευρωζώνης είναι ένα σημαντικό βήμα δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. δεν αρκεί όμως ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων χρειάζεται να καταπολεμήσουμε τα αίτια στη ρίζα τους όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάνουμε λάθο και υπονομεύουμε το κοινό μα μέλλον και το μέλλον των επόμενων γενιών δίνοντας έμφαση μόνο στην άμεση δημοσιονομική εξυγίανση και υποτιμώντας τι επιπτώσεις στην ανάπτυξη την απασχόληση και στις βασικές δομές του κράτους πρόνοιας που μας πήρε μερικές δεκαετίες για να το οικοδομήσουμε. κύριε επίτροπε οι προτάσεις που παρουσιάσατε στις 12 μαΐου για την ενίσχυση του οικονομικού συντονισμού μπορούν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ευρώπης περισσότερο συνεκτικής με λιγότερες μακροοικονομικές ανισορροπίες υπό δύο προϋποθέσεις ότι δεν θα περιοριστούν στην απαρέκκλητη εφαρμογή του συμφώνου Σταθερότητα και ανάπτυξης αλλά θα ενσωματώσουν με ουσιαστικό τρόπο εξειδικευμένους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής. 2020. ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ράγκελ για δύο, <coughs> για δύο λεπτά με συγχωρείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι από το ΕΛΚ έδωσαν μια εικόνα αρκετά πλήρη της κατάστασης. Πιστεύω ότι τώρα θα πρέπει να γίνει μια αναφορά και στο ρόλο των κρατών μελών, των εθνικών κρατών. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν εδώ ένα ρόλο να διαδραματίσουν. Υπό την έννοια ότι θα πρέπει να επιβάλλουν στα κράτη τους τις ε, απαιτήσει που χρειάζονται και τις προποθέσει ώστε το ενιαίο νόμισμα να μπορέσει να ενισχυθεί και το σχέδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης να περατωθεί. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το δικό μας κόμμα το κόμμα που συνδέεται με το ΕΛΚ στην Πορτογαλία υποβάλλει αυτές τις προτάσεις στην κυβέρνηση διότι θεωρούμε ότι εδώ και 15 χρόνια η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Πορτογαλίας που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τα σφάλματα των προηγουμένων πρέπει να αναλάβει όμως και την επανόρθωσή τους και είναι μεταξύ των δικών μας ρόλων να φροντίσουμε για τη διόρθωση των σφαλμάτων αυτών. Το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και κριτική στην πορτογαλική κυβέρνηση. Πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες. Πρέπει όχι να αυξήσουμε τους φόρους για να περιοριστεί το έλλειμμα, αλλά να περιοριστούν οι δαπάνες. Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να έχει την τόλμη να αναλάβει μέτρα τα οποία θα μετριάσουν τι δαπάνε, άρα και το έλλειμμα, άρα και το δημόσιο χρέο. Αυτό ισχύει και για την Πορτογαλία και για άλλα κράτη, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε μια δυσχερή κατάσταση. Εμεί, ω ευρωβουλευτέ, έχουμε την ευθύνη και στι δικέ μα χώρε να φροντίσουμε να υποστηρίξουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενισχυθεί κατά επέκταση και το ευρώ και να κάνουμε ένα βήμα προόδου για την ε, Οικονομική Ένωση με το ευρώ. Το κοινό όραμα λοιπόν του ΕΛΚ θα πρέπει να προωθηθεί από εμά. Κριτικάρουμε λοιπόν τι κυβερνήσει που δεν έχουν στι χώρε του το θάρρο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Ο κύριος Φάρμ για 1,5 λεπτό. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Η κρίση έχει επιπτώσεις και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τα μεγάλα στρατηγικά έργα της Ευρώπης 2020 θα χρειαστεί για να γίνουν να υπάρξει σοβαρότατος έλεγχος των δαπανών. Μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές χώρες μέλη πλέον που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση με τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα. Από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει με τη λήψη μέτρων που είναι σημαντικά για να οδηγήσουν στην ανάκαμψη των χωρών μελών. Για το λόγο αυτό, ο κοινοτικός προϋπολογισμός πρέπει να ρίξει το βάρος του ιδιαίτερα στους τομείς εκείνους όπου μπορεί να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έτσι ώστε ο προϋπολογισμός αυτός να αποδώσει και η Ένωση να ενισχυθεί. Όμως οι χώρες μέλη, εάν αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα καθήκοντα, πρέπει να την εξοπλίσουν και με περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα. Για παράδειγμα στην έρευνα. Για τον λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την οικονομική πολιτική να τηρήσουμε επικοδομητική στάση και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό για τις συζητήσεις για τη δημοσιονομική προοπτική μετά το έτος 2013. Εάν δεν το πράξουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινά μέτρα υπέρ της απασχόλησης. Κύριε Πρόεδρε, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής θα ήθελα να επαναλάβω και στην αίθουσα αυτή κάτι που έχω πει δημόσια από την αρχή και στην Ελλάδα και να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη βοήθεια που έλαβε η χώρα μου από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ο οποίος σε συνδυασμό με σκληρά αλλά ως επί το πλείστον αναπόφευκτα μέτρα απέτρεψε το άμεσο αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η ελληνική οικονομία. θα ήταν χρήσιμο αν ο μηχανισμός για την ελλάδα είχε υιοθετηθεί με την ταχύτητα που προχώρησε ο μηχανισμό στήριξη των άλλων οικονομιών όταν επιτέλου η ευρώπη συνειδητοποίησε του κινδύνου που όλοι διατρέχουμε. είναι η πρώτη φορά σήμερα που βλέπω και στο κοινοβούλιο και στους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς πραγματική αποφασιστικότητα να δούμε με αμεσότητα και ρεαλισμό τα πραγματικά οικονομικά αδιέξοδα της ευρώπης. γιατί όμως οδηγηθήκαμε εδώ; ο κύριος λόγος είναι ότι ξοδεύαμε περισσότερα από ό,τι διαθέταμε και στέλαμε το λογαριασμό στο μέλλον. ξοδεύαμε όταν δεν είχαμε κρίση ξοδεύαμε στη διάρκεια της κρίσης ξοδεύουμε τώρα που βγαίνουμε από την κρίση. όποιος θέλει να μάθει τι παθαίνει κάποιος που ξοδεύει συνεχώς χρήματα που δεν διαθέτει δεν έχει παρά να έρθει στην ελλάδα. το ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο και οι άλλοι θεσμοί που προτείνονται στο υποδιαπραγμάτευση ψήφισμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. όμως το ταμείο για να προσφέρει πραγματικά κίνητρα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το απόλυτο ύψος του χρέους και του ελλείμματος αλλά και την ταχύτητα μείωσης του χρέους και του ελλείμματο κύριοι συνάδελφοι το πραγματικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουν ανακαλύψει τον καπιταλισμό και αυτό το λέω και προς την αριστερή πτέρυγα τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο που ζουν με 200 ευρώ το μήνα και διεκδικούν τους παγκόσμιους πόρους και αγορές από εμάς τους πλουσίους που ζούμε με 2.000 ευρώ το μήνα. Δεν έχουμε πια στη Δύση το μονοπόλιο του καπιταλισμού επί του οποίου οικοδομήθηκε το παλιό ευρωπαϊκό μοντέλο. Αν δεν αλλάξουμε αν δεν τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα με διαρθρωτικές αλλαγές ανταγωνιστικότητα και καινοτομία απλώς θα ζήσουμε φτωχότερα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χούμπνερ για δύο λεπτά. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σαφώς η τωρινή κρίση είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέτρα που ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν εφαρμοστεί. Η αρμοδιότητα των ηθινόντων και των πολιτικών σχεδιαστών είναι να αναλάβουν δράση σε δύο επίπεδα για να ανακτήσουν την ισορροπία που έχει καταστραφεί από την αποτυχία των αγορών αλλά και να επανορθώσουν τι κυβερνητικέ πολιτικέ. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει όμω. Πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα και με ποια πολιτικά μέτρα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιστρέψουν στον προηγούμενο ρυθμό ανάπτυξή του. Ε, ο κανονισμό που προτείνεται δεν είναι ε, εγγύηση για το να ξεπεράσουμε την σημερινή κρίση. Επιλέξαμε να, να αναλάβουμε περισσότερα μέτρα. Όμω αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από περισσότερη απλούστευση για να μειωθεί η πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι σημερινέ φορολογικέ και νομισματικέ πολιτικέ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις απαραίτητες διευθυντικές πολιτικές. Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπου έχουμε χρέη και ελλείμματα από πάρα πολλά χρόνια, τα οποία ε, ο πληθωρισμός, τα κοινωνικά προβλήματα, η χαμηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δράσουμε για να γίνουν περισσότερα. Η αποτελεσματικότητα χρήση των δημοσίων κονδυλίων και των ευρωπαϊκών και των κρατικών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Ε, το ρυθμιστικό περιβάλλον που είναι φιλικό προ τι επιχειρήσει, οι φόροι που να μην επιφέρουν στρεβλώσει, τα κυβερνητικά μέτρα που να επιτρέπουν την ανάπτυξη, η μη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα σύστημα που να επιζητά την καινοτομία και να αποφεύγει το χρέο, όλα αυτά είναι βασικά μέτρα τα οποία πρέπει να επιδιωχθούν ώστε να επιδιώξουμε την αύξηση, την ανταγωνιστικότητα. Ε, στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μια στρατηγική η οποία να έχει αυστηρή φορολογική προσέγγιση, αλλά κυρίω να επικεντρωθεί στην καινοτομία, ώστε να επιδιώξουμε την οικονομική ανάπτυξη και αύξηση με έναν τρόπο βιώσιμο. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε και πάλι το στατικό ρόλο που μα αρμόζει και να προτείνουμε μεγάλε ευρωπαϊκέ λύσει και στου πολίτε και στι αγορέ. Το χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Μίτσελ για δύο λεπτά. Thank Mr. President. Uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θεωρώ δεδομένο ότι τα κυρίαρχα κράτη θα πρέπει να είναι υπόλογα για τι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει και για του στόχου που έχουν επιδιωχθεί και έχουν ε, δεσμευτεί να αναλάβουν. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι περαιτέρω δράσει μπορούν να συνεισφέρουν, ε, στη, να έχουν δημιουργήσει μάλλον τα σημερινά προβλήματα. Τη δεκαετία του 30 ο προστατευτισμό ε, είχε οδηγήσει σε ένταση τη ύφεση. Όμω στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προσχεθεί αλληλεγγύη και θεσμική αποτελεσματικότητα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, στηρίζουν τα κράτη-μέλη. Ε, ήδη τα αποτελέσματά μα ήταν εντυπωσιακά, δεδομένων των 27 κρατών μελών που συμμετέχουν και των 16 μελών τη Ευρωζώνη. Όμω, ε, τα θεσμικά μα όργανα πρέπει να συνεργάζονται εκτό από την Αγγλική Τράπεζα και με όλου του υπόλοιπου παγκοσμίω στην Ιαπωνία και στι ΗΠΑ. Οι αποκαλούμενε όμω αγορέ, οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, δεν έχουν ε, εξαλείψει την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τα βήματα που έχουν γίνει ως εδώ. Οι ελεύθερες αγορές είναι ένας στόχος, όμως οι αγορές μας είναι πραγματικά ελεύθερες σήμερα. Ε, επηρεάζουν στο να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να περάσουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχει μεγάλη καχυποψία ότι δεν μπορούμε ως κυρίαρχα κράτη να κερδίσουμε χωρίς αυτήν την ανάληψη μέτρων. Ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας και δεν θα προωθήσουμε την ημερήσια διαταξή μας, εάν δεν χρησιμοποιούμε τις αγορές για τους σωστού σκοπούς. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στο μέλλον της Ευρώπης να μην είναι το δολάριο το μόνο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αγορά πετρελαίου, λόγου χάρη. Θα πρέπει να μην καταστραφούν τα κυρίαρχα κράτη των δικαιωμάτων ε, με λανθασμένα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι ακριβώ συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παναλαμβάνω από τα κράτη-μέλη, πρέπει να δείξουν πειθαρχία. Και το κάτω μέλο από το οποίο εγώ προέρχομαι, αυτό έχει ήδη επιδιωχθεί. Όμω πρέπει μεταξύ των κρατών μελών να υπάρχει μια κοινή πολιτική, να μην υπάρχουν καθυστερήσει και η δραστηριότητα των αγορών να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει και ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου και τη Επιτροπή όταν δεν θα έχουμε ε, πείσει του πολίτε στο παρελθόν, τι θα κάνουμε τώρα για να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική για το 2020 είναι εξαιρετικά σημαντική. Σήμερα περισσότερο από ποτέ μέσα στα πλαίσια δηλαδή της κρίσεως. Η κρίση η οποία θέτει ερωτήματα και έχει αρνητικές συνέπειες. Η μελέτη των ερωτημάτων αυτών είναι απαραίτητο να γίνει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μειωθεί το κύρος του ευρώ πρέπει να πράξουμε πάνω το δυνατό για να διατηρηθεί το κύρος και αξιοπιστία του ευρώ και της Ένωσης. Οι χώρες που ανήκουν στην ζώνη ευρώ θεωρούν το ευρώ επιτυχία. Πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε και οι χώρες αυτές δηλαδή με κάθε τρόπο στην υποστήριξη του νομίσματος. Η κρίση μπορεί να έχει και πολιτικούς αντικτύπους. Θα ενισχυθεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στην Ευρώπη, ο ευρωσκεπτικισμός δηλαδή, και ο κόσμος θα χάσει την εμπιστοσύνη του. Οι χώρες που ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στη, χώρα, στη ζώνη ευρώ πρέπει να ενισχυθούν για να μπορέσουν να το πράξουν. Η ατζέντα του 2020 πρέπει να λάβει υπόψη και τα θέματα ασφάλειας της ενέργειας. Πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικέ πηγές, πηγές προμήθειας ενέργειας και βεβαίως να λάβουμε υπόψη και τις αναλλακτικέ ενέργειες για το μέλλον. Για να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα την ενέργεια που χρειαζόμαστε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλες τις πηγές ενέργειας όπως είπα προηγουμένως, καθώς επίσης βέβαια και την, ε, τις εκπομπές διοξιδιών του άνθρακος και άλλων αερίων του θερμοκηπίου Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν μέσα στη στρατηγική για το 2020. Πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμό όλων των τομέων, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί η Οικονομική Ένωση. Σα ευχαριστώ. Τα μέτρα που πρότειναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι ευπρόσδεκτα και μάλιστα αν είχαν ληφθεί πιο έγκαιρα, ίσως είχαν αποτρέψει ένα σημαντικό τμήμα της κρίσης. Η έλλειψη της οικονομικής διακυβέρνησης μας οδήγησε σε λήψη αποφάσεων ερήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς διαβούλευση μαζί του. Επίσης δεν υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί για τη συνέχιση αυτών των μέτρων. Πέρυσι τεράστια κονδύλια και κεφάλαια δόθηκαν στις τράπεζες που ήταν απαραίτητα ε, για τη διάσωσή του. Παρ' όλα αυτά η διάσωση των τραπεζών δεν βοήθησε την υπόλοιπη οικονομία. Το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη δεν τηρήθηκε. Τα δημόσια ελλείμματα διονγκώθηκαν και τα κράτη-μέλη για παρόμοιες καταστάσεις έλαβαν πολύ διαφορετικά μέτρα. Κάποιες κυβερνήσεις ε, αποφάσισαν να πούν την αλήθεια στους πολίτες τους και να θετήσουν μέτρα λιτότητας, ενώ άλλες κυβερνήσεις δεν έκαναν κάτι τέτοιο, κάτι που οδήγησε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα και συνέπειες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλες οι κυβερνήσεις είναι συνυπεύθυνες για την κρίση. Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε. Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε με τη φορολογία θα πρέπει να ανακτήσουμε την ε, φορολογική μας ε, σταθερότητα. Χρειαζόμαστε ένα νέο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και μία δημοσιονομική σταθεροποίηση. Φυσικά θέλουμε και μηχανισμούς συνέχισης και ανάκαμψης ε, της υγείας των δημοσιονομικών μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική οικονομική διακυβέρνηση προς όφελος όλων των κρατών μελών. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο Επιτροπή. Ε, θα αφιερώσουν πολύ λόγο στη δευτερολογία τους. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να υπερβούμε το, τους αυστηρούς κανόνες του Catch Θα προτιμούσα, επειδή είναι πολύ εγγεγραμμένοι στο κατάλογο, να έχουν ένα λεπτό ο καθένας. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, θα ακολουθήσω τους κανόνες. Καλωσορίζω την Ισπανική κυβέρνηση για το επικοδομητικό σύστημα που μας παρουσίασε για την επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Σε σχέση με τα σχόλιά σας για την ανταπόκριση θα πρέπει να δούμε κατά πόσον βρίσκεται σε τέλμα το ευρωπαϊκό σύστημα σε σχέση με την άμεση ανταπόκριση. Να δούμε δηλαδή εάν τα κράτη-μέλη μπορούσαν να είχαν αντιδράσει με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν ε, ξέσπασε η τραπεζική κρίση. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στην τωρινή κρίση, λόγω χάρη. Και τέλο, η Επιτροπή ε, αναζητά τέσσερι πυλώνε για τη σημερινή στρατηγική τη. Νομίζω η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τον ίδιο το δικό τη ρόλο στην σημερινή κρίση. Διότι το Σύμφωνο Ανάπτυξη και Σταθερότητα ήταν ίσω μια ήπια προσέγγιση ω τώρα, η οποία όμω δεν έχει δώσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πολλοί έχουν πει εδώ και εμεί ότι ίσω δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημερινό πρόβλημα εάν είχατε ήδη αξιοποιήσει τι εξουσίε που προβλέπονται για σά πλήρω. Για ένα λεπτό această perioadă de criză economică, strategia Η περίοδος αυτή της οικονομικής κρίσης και η στρατηγική Ευρώπη 2020 δημιουργούν ταυτόχρονα και προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Θα μπορούσαν να μας δώσουν ενάυσματα για να υποστηρίξουμε τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα. Και μάλιστα οι αρχές της αλληλεγγύης και της προσαρμοστικότητας θα πρέπει να πριτανεύσουν στα πλαίσια αυτών των μεταρρυθμίσεων. Α μην ξεχνούμε και τη θεμελιώδη σημασία των διαρθρωτικών ταμείων στον περιορισμό των ε, μεγάλων διαφορών μεταξύ των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα είναι προφανέ ότι οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν αυτόματα να μετατραπούν σε εθνικούς στόχους. Θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Η ρουμανική κυβέρνηση συγκρότησε μία ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου για τη θέσπιση των εθνικών στόχων και το συντονισμό του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος οι συμπεριφορέ των αγορών αλλά και των τραπεζών μοιάζουν με αγέλη λύκων όπω είπε χαρακτηριστικά ο σουηδό υπουργό οικονομικών μια αγέλη λύκων έτοιμη να κατασπαράξει τα αδύναμα οικονομικά κράτη. πρώτο θύμα η ελλάδα ακολουθεί η ισπανία και η πορτογαλία. είδαμε στην περίπτωση τη ελλάδα του κερδοσκόπου να χτυπούν ανελαίητα και την κοινοτική αλληλεγγύη να εκδηλώνεται πολύ πολύ αργά και με σκληρότατου όρου που εξαναγκάζουν τον ελληνικό λαό σε δυσβάσταχτε θυσίε και δικαιολογημένε απεργίε φαίνεται ότι η διεθνή οικονομική κρίση έχει τώρα πρωταγωνιστέ τα κράτη και όχι τι τράπεζε. από τα παθήματα α πάρουμε τα μαθήματα. η ευρωπαϊκή ένωση χρειάζεται περισσότερη κοινοτική αλληλεγγύη εποπτεία καλύτερη του χρηματοπιστωτικού συστήματο, ενισχυμένη εθνική συμμόρφωση με το σύμφωνο σταθερότητα, αυξημένο συντονισμό για τη δημοσιονομική πολιτική πρόληψη των ανισορροπιών στην ανταγωνιστικότητα. οι λαοί τη Ευρώπη, απαιτούν μια ευρώπη πιο ανθρώπινη με Λιγότερε ανισότητες ανάμεσα στα κράτη μέλη. είναι η ώρα τώρα για ένα πιο ρεαλιστικό και ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή ένωση του 2020 που να αφογκράζεται τις προκλήσεις των καιρών. Ο κύριος Σμιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη αλληλεγγύη και όχι εθνικισμό, όχι προστατευτισμό. Περί αυτού πρόκειται. Μα το έχει διδάξει η ιστορία αυτό. Βρίσκω δύσκολο να αντιληφθώ πώς έδρασαν και πώς αντέδρασαν οι Υπουργοί Οικονομικών σε σχέση με τον προπολογισμό. Δεν μπορούμε πλέον να αρκεστούμε στο να ελέγχουν οι Υπουργοί Οικονομικών τις άλλες χώρες και όχι τις δικές τους. Όλες οι χώρες εξαρτώνται από τις άλλες. Και η Σουηδική κυβέρνηση, κύριε Όλι Ρεν, και η Φιλανδία διδάχθηκε ήδη από την κρίση των, της δεκαετίας του 90. Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η πολιτική αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ε, καταστάσεως. Άλλο βήμα θα πρέπει να είναι η καταβολή προσπαθειών για να αλλάξει η κατανομή έργου των χωρών. Ένα μέγα μέρος των πληθυσμών απασχολούνται σε μη παραγωγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στην διοίκηση. Δεν είναι δυνατόν οι υπόλοιποι να εργάζονται σκληρά για να ταΐζουν τους γραφειοκράτες. Κύριε Επίτροπε, κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ασία. Εκεί ίσως να μην υπάρχουν τόσα πολλά πανεπιστήμια όσο σε εμάς, αλλά η διοίκηση επίσης δεν είναι τόσο πολυάριθμη. Και γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί μια φυσική άμυλα, ένας φυσικός ανταγωνισμός. Η απλοποίηση των κανόνων για τις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης. Για ένα λεπτό. economic crisis is not a temporary... Ε, οικονομική κρίση δεν είναι μια προσωρινή ασθένεια από την οποία τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναρρώσουν άμεσα για να ανακτήσουν την υγεία τους. Υπάρχουν μακροπρόθεσμα προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Ε, μέλη της. Το ενιαίο νόμισμα ε, για τα 16 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και για τα 27 υπόλοιπα ε, συνολικά κράτη ε, υποθέτει ότι θα είναι εύρωστες πάντοτε οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Ε, βεβαίως το νόμισμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το, την κατάσταση της υγείας των ίδιων των κρατικών οικονομιών. Όμως υπάρχει υπάρχει και η παγκοσμιοποίηση την οποία έχουν θετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Αυτό ίσω είναι μια συνταγή καταστροφή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στου εργαζόμενου από χώρε που απαιτούν χαμηλού μισθού να έρχονται στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε τα αγαθά να τα ε, κάνουμε ανταγωνιστικά όταν παράγονται με τέτοιου χαμηλού μισθού και όταν ε, οι δικοί μας εργαζόμενοι έχουν τον ανταγωνισμό των ε, μεταναστευόντων εργαζομένων ή όταν οι επιχειρήσεις μας μετατοπίζονται στον τρίτο κόσμο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Ρεν, τον Επίτροπο κύριο Ρεν, για τα καλά του λόγια και για τα καλά λόγια που είπε για την Εστονία και την ένταξή της στην ζώνη ευρώ. με 7,5% του ΑΕΠ η Εστονία δεν πρόκειται να συμβάλλει στην αύξηση του μέσου όρου του ευρωπαϊκού ελλείμματος. Είναι θετικό παράδειγμα η χώρα μου. Και είναι ενθαρρυντικό μήνυμα και προς την Λιθουανία που θα τους πείσει, θα πείσει τους Λιθουανούς ότι έχει νόημα να καταβάλουν προσπάθειες και ότι όλες οι αιτήσει των ένταξης των χωρών θα κριθούν με τα ίδια κριτήρια. Δεν είναι απλώς προνόμιο η δυνατότητα ένταξη στη ζώνη ευρώ. Σημαίνει και ανάληψη δεσμεύσεων και ανάληψη υποχρεώσεων τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητα. Εγώ πάντω είμαι βέβαιο ότι είναι η σωστή απόφαση. Θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώ μια ευκαιρία, αλλά ως μια σημαντική δυνατότητα να προωθήσουμε το κοινο, τους κοινούς μας στόχους. Ο κύριος ε, Μπέγκε για ένα λεπτό. Herr Böge, ein Minuten. Äh, ο κύριος, ησυχία, no. Äh, η κυρία ε, Γιαλοβιέσκα, για ένα λεπτό. Dziękuję, panie przewodniczący Ευχαριστώ. Η σημερινή συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιώδη σημασία γιατί αφορά την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίηση για το σύνολο της οικονομική κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα από εμά δεν θα πρέπει να έχει αφιβολία ότι μια υποπτία Συγγνώμη που σα διακόπτω, λέει ο αλλά πάτε πολύ γρήγορα για του διερμηνείς. Επιβραδύνετε παρακαλώ λίγο το αριθμό σα. Πιστεύω ότι κανένα από εμά δεν θα πρέπει να έχει αμφιβολία ότι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των δημοσίων οικονομικών και η θέσπιση των προπολογισμών καθώ και των σχεδίων μεταρρύθμιση στα κράτη-μέλη σε έγκαιρο στάδιο είναι σημαντικά μέτρα για την επίλυση τη κρίση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η εφαρμογή των αρχών του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και δημοσιονομική αλλά και μακροοικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κατονομασία των ενόχων είναι σημαντική για να αποκαταστήσουμε αυτή την εξυγίαση των οικονομικών και επίσης να θεσπίσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να τις συνοδεύσουμε από οικονομικές κυρώσεις. Γιατί πολλές χώρες ε, διανύουν ε, ε, δύσκολη οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε με υπεύθυνο τρόπο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσα σε μια κρίση το ένστικτό μας είναι πρώτα να ψάξουμε να βρούμε άλλους υπεύθυνου. Βλέπουμε επίσης να αυξάνεται, να εντείνεται ο εθνικισμός και ο προστατευτισμός αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά σωστά. Όσο περισσότερο δράσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και λιγότερο στο εθνικό, τόσο πιο εύκολα θα δαμάσουμε τις δυνάμεις των αγορών. Ωστόσο, ένα πράγμα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε να δακτυλοδεικτούμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα, ο ελληνικό λαό, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, οι Έλληνε πολιτικοί χρειάζονται το σεβασμό και την υποστήριξή μα γιατί προχωρούν στη λήψη πολύ δύσκολων αποφάσεων. Όπως είπε προηγουμένως ένας συνάδελφος, και η Σουηδία και η Φιλανδία είχαν παρόμοιε δύσκολε καταστάσει στι αρχέ τη δεκαετία του 1990 και πήραμε δύσκολε αποφάσει. Nice Σημειώνω ότι επειδή λέγατε πολύ ωραία πράγματα για την Ελλάδα, δεν σα διέκοψα αμέσω και σα έδωσα 8 δευτερόλεπτα παραπάνω. Ο κ. Φέντερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, στην παρούσα ε, συζήτηση μια λειτουργική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση πρέπει να εξετάσουμε πρώτα την ένταξη των βραχυπρόθεσμων μέτρων σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα όραμα. Η βασική αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς έχει ενταχθεί στην συνθήκη της Λισαβόνας. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς υπήρξε η ε, σπίθα εκείνη που ε, επέτρεψε την ανάκαμψη της ε, γερμανικής οικονομίας μετά τον πόλεμο. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια προσέγγιση με κρατικά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν το πλαίσιο για τη δημιουργία απασχόλησης. Όχι το ίδιο το κράτος να δημιουργήσει την απασχόληση, αλλά να θέσει τα πλαίσια για την δημιουργία απασχόλησης και ανταγωνισμού. Ο κύριος Σόμπερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ασχολούμαστε με τις ρίζες της, σημαντικής, της σημερινής μάλλον κρίσης. Ήταν σωστό να φτιαχτεί ένα κοινό νόμισμα και μια ε, νομισματική ένωση αλλά αμερικανικά χωρίς να υπάρχουν οι άλλες προϋποθέσεις. Βασίζεται ο γίγαντας αυτό σε πύληνα πόδια. Νομισματική ένωση, νομισματική ένωση μόνο με σκληρό νόμισμα. Δεν μπορεί η νομισματική αυτή ένωση να είναι αποκομμένη από την πραγματική οικονομία στο μέλλον. Επομένως χρειάζεται ξεκάθαρη ρύθμιση, ξεκάθαρες ρυθμίσεις κατά των κερδοσκόπων κατά των hedge funds και για το μέλλον και για το 2020. Σοβαρή φορολογική πολιτική με φορολόγηση των κερδών των τραπεζών. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Ας επιβάλλουμε λοιπόν τα πράγματα αυτά στον ε, ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης, όποιοι απατούν με ψευδή στατιστικά στοιχεία να φεύγουν από την Ευρωζώνη. Ο κύριος ε, Ρούμπικ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, η στρατηγική του 2020 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Και κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές πρέπει να εξετάσουμε πρωτίστως. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις να έχουν μια ένα ελάχιστο ίδιο κεφάλαιο της τάξης του 20% να το διαθέτουν το κεφάλαιο αυτό. Μην λησμονούμε ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης και ε, συμβάλλει στην δημιουργία του 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των χωρών. Μην τα λησμονούμε αυτά και να βάλουμε στόχους για την ενίσχυση των μικρών και μεσών επιχειρήσεων, να τα περιλάβει αυτά στο πρόγραμμά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσά, κύριε Επίτροπε, Κύριε Ρεν, σας παρακαλώ να καταβάλλετε προσπάθειες για να ενισχύσετε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Ε, ο κύριος Σουβέρ, για ένα λεπτό. Ε, Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, σήμερα Ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κρίση και μάλιστα ιδιαίτερα για την κρίση στην Ελλάδα. Και οι περισσότερες ε, συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο οργάνωσής μας στο μέλλον. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που θέλουν οπωσδήποτε να βρουν ε, ένοχο για αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να προβληματιστούμε ποιος είναι υπεύθυνο όχι μόνο μια συλλογική ευθύνη των θεσμικών οργάνων και της Ένωσης. Θα θέλαμε να ισχύσει η λογοδοσία και η απόδοση ευθυνών. Ο κύριος Αλμούνια, πρώην Επίτροπος Οικονομικών, ήταν ε, πολύ επικριτικός ε, απέναντι σε ορισμένα κράτη-μέλη στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Παρ' όλα αυτά όμως φτάσαμε στην κατάσταση της Ελλάδας. Θα ήθελα να παραιτηθεί αν δεν ε, μας εξηγήσει τον ρόλο που έπαιξε προηγουμένως. Ευχαριστώ. Μέσα σε ένα λεπτό τι να πρωτοπροράβω να πω κύριε Πρόεδρε. Είχαμε ήδη μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που οφείλεται στην έλλειψη ρύθμιση, εποπτείας και διακυβέρνηση. Τώρα με τα νέα μέτρα προσπαθούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον. Χαιρόμαστε για τα μέτρα αυτά και θα πρέπει να εφαρμόσουμε τέτοια πειθαρχία και στις κυβερνήσεις αλλά και στους ιδιώτες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε και τους οικονομικούς τρομοκράτες που είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης και τους ε, χρηματομεσίτες που εκμεταλλεύονται τις οικονομίες ε, των ε, ανθρώπων. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης σε πολιτικό επίπεδο, αλλά να πατάξουμε και την οικονομική τρομοκρατία, για να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κυρίε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Εκπρόσωπε του Συμβουλίου, μιλούμε σήμερα για μια κοινή ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ας μην ότι η αγορά από μόνη της δεν αποτελεί αξία. Οι Ευρωπαίοι δεν βρίσκονται εδώ για να εξυπηρετούν τις αγορές. Οι αγορές εξυπηρετούν, η αγορά δηλαδή εξυπηρετεί τους πολίτες, τα 500 τόσια εκατομμύρια Ευρωπαίων. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Ανάπτυξη αλλά που να συμβαδίζει με την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Χρειαζόμαστε λοιπόν για να επιτευχθεί αυτό αξιοπιστία. Ο κόσμο χρειάζεται να έχει προοπτικέ. Τι προοπτικέ θα του τι δώσουμε μόνο εάν μπορέσουμε να του υποσχεθούμε αλλά και να θέσουμε, να βάλουμε στα σκαριά και μέτρα που θα του επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην δημιουργούμενη ευημερία. Ανάπτυξη η οποία θα εξυπηρετήσει μόνο λίγου δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη του μέλλοντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, το μεγάλο πρόβλημα με την ελληνική κρίση έχει δημιουργήσει πολλή ανασφάλεια και στους υπόλοιπους συμπολίτε μας, όπως είναι φυσικό. Όπω είπαν και κάποιοι από του προηγούμενου συναδελφού, δεν είναι καλό να γίνει η Ελλάδα δακτυλοδεικτούμενη. Όμω είναι κατεπήγον επίση, και το συζητάμε εδώ και καιρό, να δούμε ποια είναι τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε και τι πρέπει να κάνει η ευρωπαϊκή πολιτική ώστε να οδεύσει προ μια κοινή οικονομική πολιτική. Πρέπει σήμερα κατεπηγόντω να προτείνουμε οικονομική διακυβέρνηση και τέτοια μέτρα. Ακούω την Επιτροπή να προτείνει να, την εξέταση των εθνικών προπολογισμών προκαταρκτικά. Νομίζω ότι εδώ το κατεπήγον είναι να δούμε τι θα κάναμε την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Όχι μόνο να εξετάζουμε του εθνικού προπολογισμού πριν την κατάρτιση του ευρωπαϊκού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι τέτοιε προτάσει σε κάθε περίπτωση θα έδειχναν τις θεσμικές ασυνέπειες που υπάρχουν, θα τις υπογράμμιζαν, αλλά και την πολυπλοκότητα. Θα επέφεραν πολυπλόκε διαδικασίε τις οποίες η Ευρώπη σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση είναι κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα και όχι η προτρή εξέταση των εθνικών προπολογισμών. Mulțumesc, domnule președinte că Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό τη πάση ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 θεσπίστηκε προκειμένου να διευκολύνει την ε, ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη δεκαετία. Βέβαια, η στρατηγική αυτή δεν δείχνει ένα σαφή δρόμο ό,τι αφορά την ανάγκη αναθεώρησης ε, μιας από τις σημαντικότερες ε, κοινέ πολιτικές που είναι η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό γιατί η γεωργία είναι ένα σημαντικό μέσο για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για το 2020. Την τελευταία στιγμή μόνο μπήκε μια μνήα της γεωργίας και γι' αυτό η γεωργία ελάχιστα αναφέρεται στο έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η στρατηγική περιλαμβάνει κάποια στοιχεία για το μέλλον τη κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά δεν τη θέτει στο επίκεντρο μιας ολοκληρωμένη και σφαιρικής προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικέ ε, ε, προκλήσεις που θα δημιουργήσουν οι κλιματικέ αλλαγέ και ο διπλασιασμό ε, τη ζήτηση σε τρόφιμα. Ο κύριος Σικέρσκι. Χρειαζόμαστε διεξοδική ανάλυση των αιτίων της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, ε, της κρίσης του ευρώ, της ελληνικής κρίσης και να αποφύγουμε τη μετάθεσή της και σε άλλες χώρες. Η χρηματοπιστωτική κρίση που μετατράπηκε σε οικονομική κρίση συνέβαλε σε αυτή την κατάσταση ή θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια ευθύνη για τα λάθη μας, της ανεμελιάς μας και της απερισκεψίας μας. Δεν είχαμε οικονομική στρατηγική και διακυβέρνηση στην Ένωση. Δεν τηρήθηκε ούτε η δημοσιονομική πειθαρχία, ούτε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πολύ συχνά οι κρατικοί προπολογισμοί ήταν άσχετοι με την πραγματικότητα. Πολλά έξοδα, λίγα έσοδα. Έδειξαν μια ανευθυνότητα μερικές ευρωπαϊκές χώρες τι έγινε με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής. Μερικές χώρες μέλη δεν επέτρεψαν την, την ε, εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους κοινοτικού τους προϋπολογισμούς. Έτσι δεν ασχοληθήκαμε με την Οικονομική Ένωση ούτε με την Νομισματική Ένωση τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Καταρχάς, εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος ε, Λόπες Γαρίδου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιάζει με παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν της ε, πολιτάρχης ευρωπαϊκής ιστορίας, μιας ε, κατάστασης όμως που στο παρελθόν την είχαμε ξεπεράσει βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι σαν αυτό που ζήσαμε στο δεύτερο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν τη λέγαμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ήταν μια παρόμοια κατάσταση καμπής όταν κατέρευσε το δίχως του Βερολίνου, όταν ε, ζήσαμε την επανένωση στην Ευρώπη, όταν δημιουργήσαμε το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και προχωρήσαμε επίσης με τη νέα συνθήκη. Αυτά κάναμε στην αρχή της νέα, του νέου αιώνα με την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας που είναι η μοναδική μας διέξοδος από μια δύσκολη στιγμή όπως η σημερινή. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι η δημαγωγία ή ο προστατευτισμός. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματική εναλλακτική λύση. Η μόνη λύση είναι να επιδιώξουμε μια Ευρώπη που θα καλύψει τα κενά και τις αδυναμίες της αδυναμίες που φάνηκαν με την ε, έλευση αυτής της σοβαρότητας κρίσης που ήταν και σχεδόν άνευ προηγουμένου για ορισμένους από εμά. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση με απορριθμισμένες αγορές, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με το παραγωγικό σύστημα εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Σήμερα μάλιστα έχουμε πολύ σοβαρέ συνέπειε αυτή τη κατάσταση και σοβαρέ κοινωνικέ συνέπειε με την ανεργία. Επίση, έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα ελλείμματα. 20 από τι 27 χώρε μέλη έχουν σοβαρότατα δημοσιονομικά ελλείμματα. Επίση, θα πρέπει να βρούμε τρόπο για να αντιμετωπίσουμε μια εμφανή αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έγκυται στην έλλειψη τη οικονομική διακυβέρνηση. Και ο τρόπο για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά δεν είναι με λιγότερη Ευρώπη, με ασθενέστερη Ευρώπη, αλλά με περισσότερη, πιο ενισχυμένη Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Μην μα λέτε ότι δεν αντιδράσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε. Και ο Επιτροπός σολιρέν, αλλά και εγώ είπαμε προηγουμένω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε στην κατάσταση αυτή. Αυτή τη στιγμή όμως οι ρυθμοί επιταχύνθηκαν ακόμη περισσότερο. Η εξελίξη είναι ακόμη πιο ραγδαίες. Γι' αυτό και θα πρέπει και η αντίδρασή μας να είναι πιο άμεση και να συμβάλλει στην επίλυση των ε, προβλημάτων που εκκρεμούν ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία τη οβούσα κρίση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας προτείνω μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Συνεργασία που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εστιαστεί σε πέντε τομείς για τους οποίους θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δραστηριότητά μας και να, την εφαρμόσουμε, να εφαρμόσουμε σωστά τα μέτρα μας. Ο πρώτο αυτό τομέα είναι η αλληλεγγύη. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στα θέματα αλληλεγγύη στη ζώνη ευρώ. Γι' αυτό και ήταν πολύ σωστή η ενίσχυση προ την Ελλάδα, ο μηχανισμό στήριξη για την Ελλάδα και πολύ εύστοχη η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τριετέ ε, αυτό ταμείο, που δεν είναι ακόμη σταθερό, για 750 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιε καταστάσει κρίση ή ενισορροπία στις, στα, δημόσια, στα οικονομικά του κράτους. Και αυτό ήταν επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που το ενέκρινε και που το πρότεινε και που το ενέκρινε στις 9 Μαΐου και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μάλιστα αυτή τη στιγμή παρεβαίνει αγοράζοντας ομόλογα κρατικά χρησιμοποιώντας φυσικά τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας και τις δυνατότητες που προσφέρει. Επίσης, εξετάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία δέσμη μέτρων για την ε, οικονομική εποπτεία. Και μάλιστα χθε το ΕΚΟΦΗΝ ενέκρινε τα μέτρα ρύθμισης για τα hedge funds. Και εγκρίθηκε η ρύθμιση αυτή. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό τη διαπραγματεύση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το σύνολο του πακέτου χρηματοπιστωτική εποπτεία. Και στο πακέτο αυτό θα ρυθμιστούν και οι οργανισμοί αξιολόγηση, γιατί και οι οργανισμοί αξιολόγησης θα υπαχθούν στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής, όπως πρότειναν ορισμένοι ευρωβουλευτές. Τρίτον, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να εγκαινιαστεί και να εγκριθεί η στρατηγική για το 2020. Μία στρατηγική που ποσοτικοποιεί τους στόχους και μεταξύ τους αναφέρει και το στόχο της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης, που μέχρι στιγμής δεν είχαν ποσοτικοποιηθεί. Η στρατηγική του 2020 προβλέπει μια διακυβέρνηση. Είναι πολύ πιο απαιτητική από τη σχεδόν ανύπαρκτη στρατηγική της Λισαβόνας, όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Φερχόφστατ. Θα έχουμε μια στρατηγική που θα χρησιμοποιεί κίνητρα και ανάβσματα για την υλοποίηση των στόχων, όπως είναι η χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων ή των διαρθρωτικών ταμείων. Τέταρτο σημαντικό σημείο για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι το πακέτο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών που υπέβαλε ο Επίτροπος Όλη Ρεν στις 12 Μαΐου. Το πακέτο αυτό εξετάστηκε χθες στο Συμβούλιο Εκοφήν είναι απαραίτητο να τηρήσουμε πιστά τις συνθήκες της Λισαβόνας, που στο άρθρο 5 της συνθήκης λειτουργίας αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα. Δεν είναι απλώς ευκταίο. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συντονίσουν τις οικονομικές τους πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης. Και δίνονται να συντονίσουν και τις κοινωνικές τους πολιτικές. Και από την άποψη αυτή, το άρθρο 136 μετά από πρώτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα πρέπει να τύχει κάποιες ευάθυνση και θα πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή και αυτών των μέτρων. Επίση, θα πρέπει να επιταχύνουμε τη συζήτηση και τη λήψη απόφαση στους G20 για την ε, θέσπιση φόρου για τις ε, διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Όλα αυτά τα σημεία, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικά, αυτά τα πέντε σημεία, και πραγματικά θα μας δώσουν όθηση σε αυτή την προσπάθεια για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Και ελπίζω να τύχουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα μέτρα και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν να ληφθεί υπόψη για τα σημεία αυτά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, δεν μπορούμε να περιμένουμε για πολύ ακόμη. Και η ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ. Και όταν μιλώ για ενότητα, δεν εννοώ ενότητα και ομόνια μεταξύ των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ενότητα μεταξύ των θεσμικών οργάνων, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεσμικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεσμικό όργανο και το Συμβούλιο είναι θεσμικό όργανο. Και το Συμβούλιο είναι θεσμικό όργανο, επαναλαμβάνω. Και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ του, ώστε να δοθεί αυτή η όθηση προ την οικονομική διακυβέρνηση. Και στην επίλυση αυτών των φλεγών των προβλημάτων ώστε να αντιδράσουμε και να ξεκινήσουμε μια νέα φάση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι επωφελής για τους πολίτες που αυτό περιμένουν από εμά. Δεν περιμένουν τίποτα άλλο. Αυτό μόνο να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα και να ξεπεράσουμε την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος εξ ονόματος της Επιτροπής, ε, ο κύριος Όλι Ρεν. Ε, Commissioner, the votes will take place η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 12 και 10 κύριε Επίτροπε. Την καθυστερήσαμε λοιπόν λίγο ώστε να έχετε το χρόνο που χρειάζεστε για να ομιλήσετε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την πολύ σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση που απηχεί τη σοβαρότητα της καταστάσεως που αντιμετωπίζουμε ως Ευρώπη. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι Εκτιμώ την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης, άκουσα προσεκτικά τον κύριο Λόπες Καρίδο και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ισπανική Προεδρία για την υποστήριξή της και για την εξαιρετική συνεργασία που μας προσέφερε και σε αυτό το θέμα αλλά και σε άλλα. Συμφωνώ με όσους εξημών ζήτησαν οικονομική ένωση συμπληρωματική της νομισματικής. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Και αυτό είναι το κρίσιμο δίδαγμα που πρέπει να διδαχθούμε από την κρίση. Τρία πράγματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρώτα, να συνεχίσουμε την αμεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της κρίσης και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αποφύγαμε μια κρίση, μια πτώχευση αλλά Lehman Brothers σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε με επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα για να διαφυλάξουμε την δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρώπη και την έθραστη ακόμα οικονομική ανάκαμψη στην Ήπειρό μας. Δεύτερο, πρέπει να επιταχύνουμε και να εντείνουμε και να ολοκληρώσουμε την οικονομική μεταρρύθμιση των αγορών για το short selling, για τους οργανισμούς αξιολόγησης των οικονομιών και ούτω καθεξής. Είναι πολύ καλύτερο αυτά να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα το δυνατόν ταχύτερο. Πρέπει να δημιουργήσουμε πλαίσιο διόρθωσης του συστήματος των δημοσιονομικών αγορών και εδώ συμφωνώ με την κυρία Γιάκο Σάρη και με τον κύριο Σφόμποντα η αγορά μπορεί να είναι καλός υπηρέτης αλλά είναι κακό αφεντικό και πρέπει να εργαστούμε στη βάση της ιδέας μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τις αγορές. Για να ολοκληρώσουμε δηλαδή την μεταρρύθμιση. Τέλος, τρίτον δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, να ενισχύσουμε την σταθερότητα, δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με δημοσιονομική επισκόπηση, με την θέσπιση κυρώσεων και με κανόνες, όπως είπε και ο κύριος Κάρας, και πρέπει επίσης, διακόπτει ο Πρόεδρος, με συγχωρείτε κύριε Επιτροπέ, με, με συγχωρείτε κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής συζητήσεως σας παρακαλώ λοιπόν να διακόψετε τις συζητήσεις μέσα στην αίθουσα και να δείξετε σεβασμό στον Επίτροπο. Έχει το λόγο κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω συνηθίσει στον θόρυβο αυτό, αλλά όντω ε, θα εκτιμούσα αν δείχνατε κάποιο ενδιαφέρον για τα όσα λέω. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες αμεσοπρόθεσμης λύσης της κρίσης καθώς επίσης και μια πιο μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της αγοράς και ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτή, αυτά είναι τα τρία βασικά καθήκοντα που πρέπει να μας απασχολήσουν το δυνατόν συντομότερο. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρινέσκου, εξάλλου, που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά είναι και περισσότερα από ό,τι μπορούσε κανείς να αναμένει προεξαμήνου. η ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης έχει μόνο 10 σελίδες. Φαίνεται να είναι λίγες, αλλά είναι πλήρης συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Είναι πραγματικά heavy stuff και είναι αυτά που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη και θα υποβάλουμε σύντομα και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία και θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Βερχόφστατ είπε Ας μην περιμένουμε την ομάδα ειδικών καθηκόντων, την Task Force. Εμείς συμβάλαμε αποφασιστικά στο έργο της Task Force, της οποίας προεδρεύει ο κ. Βαν Ρόμποϊ. Θα κάνουμε όμως και χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας μας και σύντομα θα υποβάλουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης το αυτή είναι η ουσία της κοινοτικής μεθόδου και αυτό ζητήσατε και εσείς σήμερα και σωστά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση. Είναι απαραίτητο τώρα να προχωρήσουμε στην, λήψη αυτών, στην ανάληψη μάλλον αυτών των πρωτοβουλειών. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία των θεσμικών οργάνων για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε παρήγαγε τα βέλτιστα αποτελέσματά της όταν υπήρξε συμμαχία των θεσμικών οργάνων. Βασίζομαι λοιπόν στην υποστήριξή σας και είναι σημαντικό στην προσπάθεια αυτή να συμβάλλουν και τα εθνικά κοινοβούλια σε μια ολιστική αντιμετώπιση όπως είπε η κυρία Ουλάρτ Πιο σημαντικό απ' όλα είναι το εξή. Θυμηθείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βοηθήσει όλους μας να δράσουμε ταχύτερα και με αποφασιστικότητα. Παρακαλώ λοιπόν βγείτε να πείσετε τους ψηφοφόρους σας και βοηθήστε μας να πείσουμε την Προεδρία, όχι μόνο την Ισπανική Προεδρία η οποία έχει την πεποίθηση αυτή, αλλά και τις άλλες, και κάντε να ακουστεί η φωνή σας. Αναμένω από εσά να λάβετε ισχυρές θέσεις και να λάβετε τις απαραίτητες αποφάσεις για την Ευρώπη του 2020 ήδη τούτη την περίοδο συνόδου. Χρειαζόμαστε πρόσω ολοταχώς για να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση έληξε. Σε λίγα λεπτά αρχίζουν οι ψηφοφορίες.